Εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην ακρόαση για την Παλαιστίνη. Γέφυρα για την ανάπτυξη. Με ευχαρίστηση Βλέπω ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων, πράγμα που αποδεικνύει το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για το θέμα το σημερινό. Είμαι η Κορίνα Κρέτσου, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης. Είμαι υπεύθυνη της σημερινής συνεδρίαση. Γιατί πήραμε αυτή την, πήρα αυτή την αντιπροσωπεία για δύο λόγους. Διότι πολλά λέγονται και γράφονται η Παλαιστίνη και τη Μέση Ανατολή. Πάρα πολύ αμαχύνεται, αλλά σήμερα πάνω απ' όλα θα ήθελα να εξετάσουμε το θέμα αυτό από την οπτική γωνία της ανάπτυξης. Πέραν από την πολιτική μιλούμε για ανθρώπους. Εκατομμύρια άνθρωποι, γυναίκες και παιδιά που ζουν στη Γάζα, στην Ιερουσαλήμ και στη Δυτική όχθη ζουν σε κατάσταση πραγματικής ένδυας. Για πολλούς Παλαιστινίους η πείνα, η έλλειψη ύδατος και η έλλειψη συνδικών υγιεινής είναι η καθημερινότητα. Υπάρχει μόνιμη έλλειψη νοσοκομείων, γιατρών, ε, νοσηλευτικού προσωπικού, για να μην αναφέρω τα σχολεία, τους καθηγητές. Υπάρχει ε, περιραίουσα ανεργία, ε, και δεν υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για να αναπτυχθούν επιχειρήσει για εμπορικές ε, ε, συναλλαγές. Πάνω απ' όλα όμως οι ίδιοι αυτοί πολίτες των κατεχομένων στην Παλαιστίνη είναι οι πολίτες τους οποίους αρνούνται κάποιοι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ελπίζω ότι ε, σήμερα θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα από την ανθρωπιστική πλευρά και ελπίζω ότι μιλώ εξ ονόματό σα όταν λέω ότι μας ενδιαφέρει σήμερα ιδιαίτερο στο θέμα αυτό. Πώς μπορούν οι Ισραηλοί και οι Παλαιστίνοι, οι γυναίκες και οι άντρε, τα πανεπιστήμια και οι επιχειρήσει να εργαστούν από κοινού για να ξεπεράσουν αυτές τι τρομερέ δυσκολίε και να φέρουν την ειρήνη και την ευημερία σε αυτό το τόσο δοκιμασμένο μέρο του κόσμου. Πρόκειται για μία πάρα πολύ φιλόδοξη πρόκληση, αλλά πιστεύω ότι αν δεν θέσουμε τι δύσκολε ερωτήσει, ποτέ δεν θα πάρουμε τι πραγματικέ απαντήσει. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρη αυτή η ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι δυναμικός και ενεργός υποστηρικτής της ειρήνης και της ε, εξέλιξης στην Παλαιστίνη. Με τα πάρα πολλά ψηφίσματα τα, για την δουλειά που έχουν επιτελέσει αντιπροσωπείς και επιτροπές. Ε, νωρίτερα, αυτό το μήνα, εγκρίναμε ένα ψήφισμα της έκθεσης Goldstone και η ευρωπαϊκή διάσταση βεβαίως είναι πρωταρχική σημασία όσον αφορά τα κατεχόμενα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χορήγησε μισό δις ε, ευρώ για την ανάπτυξη προγραμμάτων πέρσι. Ε, τα κονδύλια τα οποία χορηγούμε εμείς ε, καταβάλλονται για θέματα υγείας, εκπαίδευσης, για τους δημοσίους υπαλλήλους, για τις ευάλωτες οικογένειες κτλ. Πιστεύω επίσης ότι αν μπορέσει να υπάρξει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών, θα μπορέσουν να ξεπεραστούν και κάποια οικονομικά προβλήματα. Ξέρουμε ποιε είναι οι ε, επιπτώσεις της ένδυα. Οι εξτρεμιστές μεταξύ των Παλαιστινίων ε, είναι αυτοί οι οποίοι στρατολογούν νέους, ε, νέα παιδιά από την Γάζα και από το Δυτική Όκθη οι οποίοι δεν έχουν καμία επιλογή μεταξύ της ανεργίας ή της, το να συμμετάσχουν σε ένα ριζοσπαστικό κίνημα. Σήμερα λοιπόν θα κοιτάξουμε αυτό το θέμα ε, στα πλαίσια δύο διαφορετικών πάνελ που θα οργανώσουμε. Στο πρώτο έχουμε τέσσερις ομιλητές που είναι εδώ και θα ασχοληθούν με θέματα ανθρωπιστικά. 40 λεπτά και ανταλλαγή απόψεων. Στο δεύτερο πάνελ ο Τόνι Μπλερ, ο οποίος θα έρθει όσον ο θα επικεντρώσει την προσοχή του σε θέματα αναπτυξιακά και θα μας πει πώς έχουν σήμερα τα πράγματα από πολιτικής πλευράς. Το πάνελ μαζί με το πάνελ αυτό γίνεται σε συνεργασία με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και θα ανταλλάξουμε μετά διάφορες απόψεις. Η... Θα ήθελα να καλεσορίσω τους τέσσερους ομιλητές μας, τον κύριο Μαξ Χάιλαρντ, ε, τον κύριο Ντέιβιτ Σίμχα, την κυρία Μπαρμπάρα Στένσον από ε, ε, και την κυρία Χάνα από το Ερευνητικό Κέντρο Ισραήλ Παρεστίνης για θέματα ενημέρωσης που είναι ένα κοινό θεσμικό όργανο Παλαιστινίων και Ισραηλινών για την επίλυση των ε, συγκρούσεων μεταξύ Ισραηλινών Παλαιστινίων. Δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Μαξ Γκέιλαρ για 10 λεπτά. Uh, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, στο πλαίσιο αυτού του δεκάλεπτου, που είναι πολύ σύντομο, νομίζω ότι αναφέρατε ότι είμαι συντονιστή του ΟΗΕ για ανθρωπιστικές υποθέσεις και ιδίως για θέματα κατοικιών στα κατεχόμενα της Παλαιστίνης. Μπορώ να μιλήσω λοιπόν και από την αναπτυξιακή προοπτική ε, αυτός είναι και ο ρόλος μου συντονιστή του ΟΗΕ για τα θέματα των κατοικιών και από την άποψη των ανθρωπιστικών ζητημάτων ως συντονιστή σε θέματα τέτοια. Να τονίσω τρία βασικά σημεία για την κατάσταση όπως έχει στην πραγματικότητα. Πρώτα απ' όλα για το τι συμβαίνει στη Λεωρίδα της Γάζας, μετά στην Δυτική Όχθη και εδώ έχουμε και τη συνάδελφο η οποία θα αναπτύξει τόσο ή στα σχετικά θέματα, την κυρία Μπάρμπαρα Σένστον και θα σας δώσει μια πιο σφαιρική εικόνα και μετά θα κλείσω με μια πιο συνολική εικόνα για την ε, οικοδόμηση κράτους που σε ό,τι αφορά την Παλαιστίνη. Σε αυτήν την ε, ακρόαση λοιπόν πρέπει να πούμε ότι έχουμε οργανώσει την συνάντηση στην επικαιρότητα διότι θα με επισκεφθεί τα κατεχόμενα ο Μπάν Κιμούν, ο γρονιονικό γραμματέα του ΟΗΕ, ενώ πριν από λίγε μέρε είπατε εκπρόσωπο, η κυρία Άστον, βρέθηκε στην περιοχή. Μιλάμε για δύο σημαντικέ επισκέψει, ενώ ο αντίστοιχο συντονιστή ε, επισκέφθηκε την περασμένη Παρασκευή τη Μόσχα. Οπότε υπάρχει συγκέντρωση της προσοχής, κινητικότητα, πολιτικές και άλλες ανησυχίες. Δεν ξέρω αν ανέφερα και το κουαρτέτο, αλλά θα πρέπει εδώ να τονίσω ότι αυτό που επιζητά το κουαρτέτο και αυτό που επιζήτησε και στην Μόσχα είναι να συνεχίσει να ενθαρρύνει τις ε, δύο πλευρές να προσέλθουν σε διαπραγματεύσεις και να καταλήξουν σε κάποια επίλυση της όλης διαφοράς ή δυνατόν στο προσεχές μέλλον. Για τη Γάζα λοιπόν να πω ότι ο Γενικός Γραμματέας ήταν μόλις χθε εκεί και η κυρία Άστον πριν από λίγες μέρες. Πώ θα μπορούσα να περιγράψω την κατάσταση αυτή τη στιγμή στη Γάζα. Θα παρακολουθείτε όλε τι εξελίξει και τι ειδήσει. Εγώ θα χρησιμοποιούσα μια πρόταση. Τα πράγματα υποβαθμίζονται από κοινωνική και οικονομική πλευρά με σοβαρότατε ανθρωπιστικέ συνέπειε. Τι εννοώ. Και πρέπει να σα πω ότι βρίσκομαι συχνά στην ε, Γάζα εβδομάδα παραβδομάδα σχεδόν. Και ένα από τα βασικά προβλήματα είναι η τροφοδοσία σε νερό και τα υγειονομικά, οι υγειονομικές υποδομές. Η λειτουργία όλου αυτού του συστήματος και του δικτύου είναι μόλις επαρκής. Λίγοι έχουν πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό. Ενώ οι δάτινοι ορίζοντες, ε, στην, οι υδροφόροι μάλλον στην Γάζα, στις οποίες ε, επαφίενται οι κάτοικοι για το πόσιμο νερό, υποβαθμίζονται και εκείνοι συνεχώ. Αυτό συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια και όλο και χειρότερα πηγαίνει. Το, το πρόγραμμα του ΟΗΕ για τα θέματα αυτά μας λέει ότι πολύ σύντομα οι υδροφόροι αυτοί ορίζοντες θα έχουν εξαντληθεί το πολύ σε 50 χρόνια. Και επίση οι ορίζοντες αυτοί αφορούν και το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Εφόσον λοιπόν το αποχετευτικό δίκτυο και το υγειονομικό αλλά και το υδροδοτικό είναι τόσο ευάλωτα, αυτό πλήττει τον πληθυσμό. Περίπου 18 εκατομμύρια λίτρα απόβλητων που δεν έχουν ε, τύχη επεξεργασίας ε, κρύπτονται στην ε, Μεσόγειο καθημερινά. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό. Όπω επίση για του κατοίκου τη Γάζα, είδαμε ότι τα επίπεδα φτώχεια από την πλευρά του ΟΗΕ συνεχώ αυξάνονται. Από άποψη οικονομικών όρων, η Γάζα θα μπορούσε να περιγραφεί τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια μια περιοχή μεσαία τάξη και οικονομική κατάσταση. Αυτή τη στιγμή όμως έχει γίνει μια περιοχή που βασίζεται μόνο στον πόλεμο και τα έσοδα των πόλεμων. Το 80% των κατοίκων ε, της Γάζας ε, για τα μετρητά, από την άποψη των μετρητών και των τροφίμων ε, βασίζονται στην ανθρωπιστική βοήθεια σε δωρητές και τους εταίρους τους. Το επίπεδο φτώχεια είναι πολύ χαμηλό. Ένα επιχειρηματική κοινότητα στη Γάζα που θα μπορούσε να είναι κινητήριος δύναμη για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη σχεδόν έχουν εξαλειφθεί. Αυτή η επιχειρηματική κοινότητα βεβαίω κάνει ό,τι μπορεί, έχει δραστηριότητα στη Γάζα. Μόλις τις προάλλες είδα να ξαναδημιουργείται μια προσπάθεια να... για μια βιομηχανία που φτιάχνει τούβλα. Με επεξεργασία των απορριμμάτων από τα ερήπια που υπάρχουν στη Γάζα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νέε οικοδομικέ εργασίε. Υπάρχει λοιπόν κάποια υποτυπώδη ε, δραστηριότητα, αλλά σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Τώρα, με, με μια, μια κουβέντα, ποιο είναι το πρόβλημα τη γάζα, Είναι πολιορκία. Για όσου δεν το γνωρίζουν, να σα το εξηγήσω, αν δεν καταλαβαίνετε την έκταση του προβλήματο τη πολιορκία. Υπάρχει ένα τείχο που χωρίζει τη λόρδα τη Γάζα και το Ισραήλ. Δεν έχει σφραγιστεί, αλλά ουσιαστικά είναι κλεισμένο. Υπάρχει και ένα τείχος με την Αίγυπτο, που χωρίζει από την Αίγυπτο, και επίσης υπάρχει και τείχος που χωρίζει την Γάζα από τη θάλασσα, τρία μίλια από την ακτή. Πραγματικά μιλάμε λοιπόν για πολιορκία για τους κατοίκους της Γάζας, εφόσον λυνόταν η πολιορκία, θα χρειαζόταν αρκετός χρόνος να ανακάμψει η περιοχή. Απλώς να σας εξηγήσω ότι πριν από λίγα χρόνια μόλις, εκατοντάδες ε, οποροφόρα φρούτα και άλλα αγροτικά προϊόντα εξάγονταν εδώ στην Ευρώπη. Υπήρχαν τουλάχιστον 2.500 3.000 οικογένειες γεωργών στην Γάζα που έχουν αυτές τις ε, ικανότητες ακόμη. Το ίδιο και οι ψαράδες στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή, και θα κλείσω εδώ για τη Γάζα, γιατί δεν θέλω να μακρηγορήσω, το 2009 μόλις, ο ΙΕ μόνον δαπάνησε για ανθρωπιστική ανακούφιση 450 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια, μόλις το 2009. Θα μπορούσα να πω ότι πολύ λίγα από αυτά τα κονδύλια θα ήταν απαραίτητα σε κανονικές συνθήκες. Τώρα για τη δυτική όχθη να πω ότι τα πράγματα είναι τόσο περίπλοκα όσο και στην Γάζα για διαφορετικού λόγου, Θα τα ακούσετε όμως με λεπτομέρειε αυτά και από τον κύριο Μπλερ. Αλλά υπάρχουν σοβαροί περιορισμοί για τι οικονομικέ δραστηριότητε σε αυτή την περιοχή. Περιορισμοί που δεν επιτρέπουν την οικονομική ανάπτυξη. Από την άποψη τη ανθρωπιστική βοήθεια δεν θα ήταν υποκανονικέ συνθήκε απαραίτητη αλλά κινητοποιούμε τον ανάλογο μηχανισμό του ΟΗΕ και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή την περιοχή. Και σε συνεργασία με συναδέλφους από μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Και σε κάθε περίπτωση ε, στην περιοχή αυτή που κατά 60% κατέχεται από το Ισραήλ. Υπάρχουν λοιπόν και άλλα κοινωνικά προβλήματα, η φτώχεια αυξάνεται, τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στα σχολεία, δεν υπάρχουν τάξεις, δεν υπάρχουν δάσκαλοι. Δεν υπάρχουν δημοτικές υπηρεσίες σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ιερουσαλήμ, της Ανατολικής ε, Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι η τρίτη περιοχή που μας ε, αφορά. Η περιοχή μεταξύ του τείχου διαχωρισμού που ουσιαστικά απέχει λίγο από την πράσινη γραμμή. Έτσι λοιπόν η κοινότητα των Παλαιστινίων βρίσκεται ακριβώ παγιδευμένη μεταξύ του τείχου και τη πράσινη γραμμή. Υπάρχουν ε, χιλιάδε άνθρωποι που ζουν σε αυτή την περιοχή και οι καλλιεργούμενε εκτάσει κανονικά, που κανονικά καλλιεργούνταν έχουν ουσιαστικά βρεθεί φυλακισμένε κι αυτέ μεταξύ της, του τείχου και τη πράσινη γραμμή. Και Λίγα λόγια για τις προτεραιότητες ως προς την οικοδόμηση του κράτους στην ε, Παλαιστίνη και το τι κάνουν γι' αυτό οι Παλαιστινιακές αρχές. Θα θυμάστε τι ανακοινώσει και τι προτεραιότητες είχαμε αναφέρει πέρσι τον Αύγουστο ήδη. Οι Παλαιστίνοι θα πρέπει να συνεχίσουν με την οικοδόμηση και την ενδυνάμωση των θεσμικών οργάνων για το κράτος και για τα ερχόμενα χρόνια. Έχουμε περάσει ήδη από 18 μήνες προσπαθειών και πολλοί λένε ότι η στόχη αυτή ήταν φιλόδοξη και μέχρι και υπερβολική. Έχουμε όμως την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να αυξήσουμε και να εντείνουμε τους ρυθμούς για την οικοδόμηση και την ενίσχυση του κράτους. Σύντομα να σας αναφέρω τα εξής τρεις στοιχεία για την ασφάλεια στα κατεχόμενα εδάφη και τι περιοχέ που ελέγχουν οι Παλαιστίνοι, τα πράγματα πρέπει να πω ότι πάνε πολύ καλύτερα. Και ο κύριο Μπλέρη να αναφερθεί σε αυτό. Στι ε, πόλει και τι κατοικίε των Παλαιστινίων, στην Ιεριχώ και σε πολλέ άλλε πόλει, με, ασφάλειες, με δυνάμεις ασφαλείας των Παλαιστινίων που είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι, με πρόσφατη εκπαίδευση η ασφάλεια έχει γνωρίσει πολύ σημαντική ενίσχυση. Καλύτερη, καλύτερη επίπεδο λοιπόν ασφαλεία στι περιοχέ αυτέ όπου υπάρχει τέτοιο έλεγχο. Ω προ την οικοδόμηση των θεσμικών οργάνων, ο Πρωθυπουργό και ο Υπουργό Οικονομικών και άλλα μέλη τη κυβέρνηση έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν μια βάση οικονομική και φορολογική πολύ ισχυρή για να τονώσουν τα οικονομικά της περιοχής. Μάλιστα αυτόν τον καιρό υπάρχουν ε, σοβαρές ελπίδες ότι τα χρήματα που διοχετεύονται στο Παλαιστινιακό σύστημα προς όφελος του Παλαιστινιακού λαού ουσιαστικά ξέρουμε πού πηγαίνουν. Παρακολουθείτε το πώς δαπανώνται και κατά τρίτον ο Πρωθυπουργός έχει απευθυνθεί σε ιδιώτες για μικρά προγράμματα στην Δυτική Όχθη, νομίζω το 2009. Ξοδεύτηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για αυτά τα προγράμματα με οικοδόμηση σχολείων, νοσοκομείων και το καθεξής. Εδώ θα ήθελα να κλείσω εγώ τη δική μου παρέμβαση, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα σας κάνουμε ερωτήσεις και θα μας δώσετε απαντήσεις για να επεκτείνουμε, για να εμβαθύνουμε στο θέμα αυτό. Να δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Ντάβιτ Σίμα. Σας ευχαριστώ. Κυρία Κωτή. Αξιότιμοι βουλευτέ, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ε, Ανάπτυξης, αξιότιμα μέλη του πάνελ, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ σήμερα ως εκπρόσωπος της ε, επιχειρηματικής ε, κοινότητας του Ισραήλ, τα μέλη της οποίας αγωνίζονται για την ανάπτυξη και την ειρήνη στην περιοχή μας. Να τονίσω ότι δεν είμαι εκπροσώπος ε, καμίας πολιτικής οργάνωσης. Δεν κατέχω οποιαδήποτε επίσημη πολιτική θέση. Βρίσκομαι εδώ εκπροσωπώντας εκείνους που επιθυμούν και ονειρεύονται ένα καλύτερο μέλλον για την περιοχή μας. Δεν ε, ήρθαμε εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για την ιστορία. Sorry. Μια σύντομη διακοπή γιατί από το μικρόφωνο του ομιλητή. Μαζευτήκαμε λοιπόν εδώ σήμερα για να συζητήσουμε όχι την ιστορία, την αρχαία και τη σύγχρονη, αλλά για να ατενίσουμε το μέλλον. Α, έχω προβλήματα με τα αγγλικά μου, αλλά θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ. Ήρθαμε λοιπόν εδώ σήμερα για να οραματιστούμε τι μπορούν να κάνουν όλοι, όλα τα μέρη που συμμετέχουν για να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής, αξιότιμοι προσκεκλημένοι. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι υπάρχουν τρόπους, τρόποι για να πετύχουμε ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον για όλους τους κατοίκους της Μέσης Ανατολής και θα πρέπει να τονίσουμε όλα τα θέματα τα οποία ενδεχομένως να καταστήσουν αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Δεν χρειαζόμαστε σλόγγαν, δεν, χρειαζόμαστε, να, δεν χρειάζεται να ακολουθήσουμε τις πεπατημένες οδούς. Πριν ε, από ένα χρόνο κάποιοι επιχειρηματίες συμπεριλαμβανομένου και τύπου υποφαινόμενου εκπροσωπώντας διάφορες επιχειρηματικές οργανώσεις στο Ισραήλ μαζεύτηκαν και δημιούργησαν το IPCC, το Ισραηλο-Παλαιστινιακό ε, βιομηχανικό επιμελητήριο, μία μη, βιο, κερδοσκοπική οργάνωση και τα μέλη των επιχειρηματιών συμπεριλαμβανομένων της Ομοσπονδίας ε, Επιμελητηρίων της Ισραηλινής, ε, του Ισραηλινού Ιδρύματος Εξαγωγών, της, του Ισραηλινού, της Ισραηλινής Ομοσπονδίας, του Κέντρου για την Ειρήνη το Επιχειρηματικό Φόρουμ, το IPBF και πολλές άλλες οργανώσεις μας βοήθησαν και μας βοηθούν για την ε, οικοδόμηση γεφυρών. Το IPCC έχει ως στόχο να βελτιώσει τις ε, διμερείς εμπορικές ροές μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων για να προωθηθούν οι επιχειρηματικές να δημιουργηθούν ισχυρά επιχειρηματικά και κοινωνικά δίκτυα και να ενισχυθεί η αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη από την ίδρυσή του. Το επιμελητήριο έχει στεφθεί με επιτυχία και είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Τόνι Μπλερ, ο οποίος ε, παρευρέθηκε και στα εγγένεια του επιμελητηρίου μας, θα χαρεί ιδιαίτερα να ακούσει ότι καταφέραμε να περπηδήσουμε ήδη πολλά σημαντικά γραφειοκρατικά εμπόδια και να σημειώσουμε σημαντικές επιτυχίες. Επιτρέψτε μου να φέρω μερικές εξ αυτών. Να ξεκινήσω με το IPCC, την οργάνωση Ομπρέλα, που περιλαμβάνει όλες τις οργανώσεις που ανέφερα προηγουμένως η ισχυρή συνεργασία για τη βελτίωση της οικονομίας της πόλεως και της βελτίωσης της συνεργασίας με τις Ισραηλινές ε, επιχειρήσεις. Η ίδρυση του επιχειρηματικού οδηγού της Παλαιστίνης που θα αποκαλύψει σε ενδεχόμενους αγοραστές ε, τα προϊόντα και τις εταιρείες. Έγιναν ε, συναντήσεις αυτά τα χρόνια μεταξύ των επιχειρηματιών και των δύο κοινοτήτων για θέματα όπως οι μεταφορές, τα τελωνία, τα τελωνιακά πρότυπα και ούτω καθεξής. Και ξεκίνησαν και συναντήσεις μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών επιχειρηματιών. Ξεκίνησε η ιστοσελίδα του IPCC. Το... Δημιουργήθηκε μία λέσχη του IPCC το Breakfast Club. Ξεκίνησαν διάφορες δραστηριότητες από το Κέντρο για την Ειρήνη και οι νεαροί Παλαιστίνοι και οι Ισραηλινοί συμμετείχαν σε ένα κοινό εργαστήριο υπό την ηγεσία του κυρίου Νίκολα Τζάνι, εμπειρογνώμονα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η πρώτη μεγάλη κλίμακα συνάντηση Ισραηλινών και Παλαιστινίων της τελευταίας δεκαετίας ε, διοργανώθηκε στην Ιεριχώ μία ε, πόλη υπό την Παλαιστινιακή Αρχή και συμμετείχαν πάνω από 120 ηγέτες ε, οργανώσεων για την διήμερη αυτή συνάντηση. Δύο διοργανώθηκαν επίσης δύο εργαστήρια για αγροτικά θέματα. Είναι η πρώτη φορά που οι αγρότες της Γάζας συμμετείχαν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα μετά από ένα ολόκληρο χρόνο. Από την περιοχή του Τουμπάς, 25 καλλιεργητές συμμετείχαν σε μία έκθεση του στο Ισραήλ το 2010. Ο τουρισμός και ένα σχετικό φόρουμ το οποίο ονομάζεται TFOP διοργάνωσε διμερεί τέτοιε συναντήσεις μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών το 2009. Πάνω από ένα εκατομμύριο τουρίστες πέρασαν στο Ισραήλ από τη Δυτική Όχθη. Κάποιες δραστηριότητες ε, του, επιμελητηρίου ε, των Ισραηλινών. Έκθεση για τα έπιπλα, B2B. Συναντήσεις για την ανάθεση της συνεργασία στον τομέα της κλωστιφαντουργία. πολύ σημαντικός τομέας. Το επιχειρηματικό φόρουμ Ισραήλ και Παλαιστίνης, το οποίο και γνωρίζετε. Συνεργασία με την ε, Σουηδική επιχειρηματική κοινότητα. Δυστυχώ, ο κύριος Χουλέλα ήταν να παρευρεθεί εδώ σήμερα, αλλά πρέπει να προετρέψει της οργάνωσης αυτή. Το 2009 το Γραφείο Στατιστικών Στοιχείων της Παλαιστίνης ανέφερε ότι το ποσοστό επιχειρήσεων στη Δυτική Όχθη ήταν 44,4% ο ρυθμός ανάπτυξης. Αυτό καταδεικνύει ότι υπάρχει λόγος να επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία από τον Σεπτέμβριο του 2009. Γιατί το ποσοστό αυτό αναμενόταν να είναι 27% και βλέπουμε ότι υπάρχουν τέτοια project χάρη στα οποία θα οικοδομηθούν πιο πολλές γέφυρες και θα έχουμε πιο πολλές ευκαιρίες για να ξεκινήσει η ειρήνη από τα κάτω προς τα πάνω, από τις ρίζες της κοινωνίας των πολιτών, στην δική μας περίπτωση από τον λαό της Παλαιστίνης και του Ισραήλ. Και να αναφέρουμε και κάτι ακόμα εδώ, προκειμένου να έχει επικοδομητικό αντίκτυπο το οτιδήποτε, θα πρέπει να βασίζεται στην πραγματική ισότητα. Και εγώ πιστεύω ότι πολλά έχουμε να μάθουμε από τους γείτονές μας στην Παλαιστίνη χωρίς αμοιβιότητα, χωρίς ε, αμοιβαία κατανόηση και σκληρή δουλειά δεν θα πετύχουμε τίποτα. 14 δισεκατομμύρια σέκελ, 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το εμπορικό συλλογισμό μεταξύ της Παλαιστινιακής Αρχής και του Ισραήλ. Αυτό είναι γεγονός. Ένα γεγονός αδιαμφισβήτητο για το, το οποίο κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει. Ναι μεν, Πολλοί ισχυρίζονται ότι η τρέχουσα στρατηγική κατάσταση θα αποσταθεροποιήσει την ε, περιοχή και όλες αυτές οι ωραίες ιδέες δεν θα μας οδηγήσουν πουθενά. Η μοναδική μου απάντηση στα επιχειρήματα αυτά είναι ότι ούτε κι εγώ ούτε και οι συνάδελφοί μου που είμαστε όλοι πολύ αφοσιωμένοι δεν μπορούμε να κατευθύνουμε τα πολιτικά διεθνή ζητήματα τα οποία περιπλέκουν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αυτό όμως που κάνουμε και που μπορούμε να κάνουμε και που θέλουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε μια νέα πραγματικότητα στην οποία η ειρήνη, η σταθερότητα, η αμοιβαία κατανόηση θα επικρατήσουν. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι το βασικό κλειδί για το όνειρό μα είναι να συνεχίσουμε τις αμοιβαίες επιχειρήσεις μας προκειμένου να διευκολύνουμε τις προσπάθειες και των δύο κυβερνήσεων προς την ειρήνευση της περιοχής. Σας ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε, κυρία Μπάρμπαρα Σένστον τώρα. Καλησπέρα σας κύριε και κύριοι. Έρχομαι ενώπιον σας ως εκπρόσωπος της UNRWA, τον οργανισμό του ΟΗΕ για την ανακούφιση και τα έργα που αφορούν τους Παλαιστινίους πρόσφυγες. Όπως ξέρετε, ο οργανισμός αυτός πριν από 60 χρόνια άρχισε να λειτουργεί ως προσωρινός οργανισμός για να προσφέρει ανακούφιση και στήριξη στους ε, πρόσφυγες. 700.000 εκείνο τον καιρό, οι οποίοι έφυγαν από τα ιστορικά εδάφη της τότε Παλαιστίνης και έχασαν ε, το τι περιουσίε του μεταξύ του 1946 και του 1948 στον πόλεμο που δείξαν στη δημιουργία του κάτω στο Ισραήλ. Με την εντολή που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1949 και επειδή δεν υπήρξε βιώσιμη και δίκαιη λύση για το, φόρτο, για το πλήγμα που δέχτηκαν, ο οργανισμό αυτό συνεχίζει σήμερα να προσφέρει προστασία και υπηρεσίε στα 4,7 εκατομμύρια πρόσφυγε που ζουν σε πέντε κέντρα επιχειρησιακά στην Μέση Ανατολή, στη Δυτική Όφη, τη Γάζα, την Ιορδανία, το Λίβανο και τη Συρία. Ως Ω ε, πρόεδρο αυτού του οργανισμού στη Δυτική Όχθη, είναι μεγάλη μου χαρά που σήμερα βρίσκομαι μαζί σα για να συζητήσω τι προοπτικέ ανάπτυξη σε αυτή την ταραγμένη περιοχή του κόσμου. Θα ξέρετε ότι θα, ο οργανισμό μα καλύπτει τι πολλέ περιοχέ, αλλά εγώ θα επικεντρωθώ στη Δυτική Όχθη. Ξέρετε ότι στην ε, Δυτική Όχθη έχουμε σήμερα 771.000 πρόσφυγες καταγεγραμμένους, περίπου 30% του πληθυσμού αυτού ε, τον, του, του συνόλου του πληθυσμού της περιοχής που ανάγεται στα 2,3 εκατομμύρια. Ε, και αυτή τη στιγμή δίνουμε τακτικές υπηρεσίες σε περίπου 600.000 πρόσφυγες. Μεταξύ των όσων προσφέρουμε περιλαμβάνεται η υγειονομική περίθαλψη, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η ανακούφιση και κοινωνικές υπηρεσίες για τους πλέον ευάλωτους. Επίσης ε, ασχολούμαστε με την ανεργία των νέων και έχουμε ένα μικρό νοσοκομείο καθώς και ένα μικρό σχολείο. Πέρα αυτών των βασικών υπηρεσιών που προσφέρονται σε όλη την Μέση Ανατολή. Η UNRWA προσφέρει και άλλα προγράμματα κατεπίγουσας βοήθειας οι οποίε είναι απαραίτητε για τα κατεχόμενα από το 2000 στην Γάζα και στην Δυτική Όχθη και πρόσφατα και στο Λίβανο. Προσφέρεται δηλαδή προστασία, τρόφιμα, ε, μετρητά εναντιεργασίας και άλλες ε, πρωτοβουλίε για την ε, επιβίωση των προσφύγων. περίπου 500 εκατομμύρια ε, ευρώ μάλλον δολάρια ε, δαπανήθηκαν ε, φέτος για την ευρύτερη περιοχή, ενώ στη Δυτική Όχθη 140 εκατομμύρια. Έχουμε 5.000 άτομα προσωπικό που εργάζονται για την προστασία των προσφύγων. Κάποιοι από αυτούς είναι δάσκαλοι και κάποιοι από αυτούς είναι οι ίδιοι πρόσφυγες. Η κατάσταση λοιπόν σήμερα. Οι πρόσφυγε τη ε, Παλαιστίνη στη Δυτική Όχθη συνεχίζουν να ζουν μια κατάσταση ανθρωπιστική και αναπτυξιακή κρίση που ολοένα και εντείνεται, με κάποιε χλωμέ προοπτικέ ε, ανάπτυξη το 2010. Για του περισσότερου πρόσφυγε, οι οποίοι βρίσκονται μεταξύ των πλέον φτωχών και ευάλωτων Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, η κατάσταση ουσιαστικά δεν έχει μεταβληθεί. Στην ουσία είναι μάλλον ε, θολή και δύσκολη. Η ουσία τη κρίση είναι η σταθερή σταθερή στρατιωτική κατοχή τη Δυτική Όχθη. Τα στοιχεία τη κατοχή αυτή σημαίνουν την εδαφική, τον εδαφικό κατακαιρματισμό, τον περιορισμό τη στη μετακίνηση των ανθρώπων και των εμπορευμάτων, την ε, ε, τελμάτωση τη οικονομική ανάπτυξη, καθώ και την συστηματική βία και ανασφάλεια, κάτι που απειλεί τη ζωή τόσο των Παλαιστινίων όσο και όλων των κατοίκων τη Δυτική Όχθη, μεταξύ των οποίων οι πρόσφυγε. Για το 2009 φάνηκαν κάποια πρώτα δείγματα οικονομική ανάπτυξη μαζί με την ε, με την, με την ε, μεγαλύτερη δυνατότητα κυκλοφορίας εσωτερικά, καθώς ε, και τις, καλύτερε τις καλύτερες συνθήκες σε μεγάλες πόλεις. Τα δείγματα αυτά είναι ευπρόσδεκτα, αλλά είναι πολύ νωρίς για να γιορτάσουμε για τη βελτίωση αυτή. Έτσι κι αλλιώ είναι πολύ αργέ οι βελτιώσει και επικεντρωμένε σε πολύ συγκεκριμένα ε, σημεία τη περιοχή η απομάκρυνση από την ανάπτυξη συνεχίζεται. Όπως μου έλεγε ο κυβερνήτης ε, της Ναπλού ε, την περασμένη εβδομάδα, ναι, μπορούν να μετακινηθούν μέσα και έξω από την πόλη οι κάτοικοι και αναπτύσσεται κάποια οικονομική δραστηριότητα, αλλά οι αλλαγέ είναι πολύ μικρές και οι επενδυτές δεν έχουν ακόμη εμπιστοσύνη για να επιστρέψουν. Ενώ κάποια σημεία ελέγχου δεν υπάρχουν πια, υπάρχουν άλλα υπτάμενα ή προσωρινά σημεία ελέγχου δηλαδή τα αντίστοιχα οδοφράγματα. Ο κυβερνήτη έλεγε ότι η κατάσταση στι μεγαλύτερε πόλει είναι ασφαλέστερη και πιο ήρεμη και αυτό χάρη στι εντατικέ προσπάθειε των καλύτερα εκπαιδευμένων και επαγγελματικών δυνάμεων ασφαλεία των Παλαιστινίων, των PSF. Όμω εκφράζει την θλίψη του για το ότι η Ισραηλινές ε, δυνάμεις, οι ε, στρατιωτικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιδρομές τους σε κατοικημένες περιοχές, προχωρούν σε συλλήψεις και υποβαθμίζουν ε, την κατάσταση των Παλαιστινίων. Σημειώνεται το σύστημα ελέγχων, οι άδειε, οι εισβολές, οι δρόμοι με ελεγχόμενη πρόσβαση είναι ισχυροί όσο και στο παρελθόν και ουσιαστικά ριζώνουν όλο και πιο βαθιά στην περιοχή. Οι παράγοντε αυτοί οδήγησαν την Παγκόσμια Τράπεζα να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι πολύ νωρί για να μιλήσουμε για νέα οικονομική δραστηριότητα στη Δυτική Όχθη. Παρόλα αυτά φαίνεται για πρώτη φορά εδώ και χρόνια να υπάρχει θετική ανάπτυξη ΑΕΠ ε, για την ΑΕΠ για την Παλαιστίνη. Μια τάση δηλαδή προς την βιώσιμη οικονομική αύξηση. Μεγάλο μέρος της ανάπτυξης αυτής οφείλεται στις δαπάνες των δωρητών με δωρεές που σκοπό έχουν να ανακουφίσουν την, ε, τον αντίκτυπο του πολέμου τη περασμένη χρονιά στη Γάζα. Όλα αυτά μπορεί να μην διαρκέσουν. Και αναγνωρίζουμε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή έχει ένα σοβαρό έλλειμμα για τη φετινή χρονιά μπροστά τη. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα περιβάλλον το οποίο να επιτρέψει, να επιτρέψει την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και πραγματικέ εμπορικέ συναλλαγέ μεταξύ χωρών και περιοχών εντό ε, τη ε, δυτική ε, όχθη. Ε, Ακόμη και η εσωτερική κυκλοφορία και η πρόσβαση σε αγορέ ε, εκτό ε, Δυτική Όχθη στη Γάζα, στο Ισραήλ, στο Ισραήλ και αλλού δεν επιτρέπεται αρκετά. Πρέπει να απελευθερωθεί. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι μια μεγάλη αλλαγή στο καθεστώ ελέγχου και ε, περιορισμού της κυκλοφορία. Δεν είναι απλό <clears throat> να αλλάξει αυτή η τάση υποβάθμισης που έχει προκαλέσει στην Παλαιστινιακή οικονομία το, το καθεστώς πολιορκίας. Ήδη από το 1999 ε, το κατακεφαλήν ΑΕΠ έχει πέσει στο 1 τρίτο τη φετινή χρονιά παρά την περιορισμένη ανάπτυξη. Το θέμα λοιπόν είναι τι θα γίνει με την επιβίωση των Παλαιστινίων, ιδίω των προσφύγων. Τα επίπεδα φτώχεια παραμένουν πολύ ψηλά μεταξύ των προσφύγων και τα ποσοστά ανεργία επίση προκαλούν ε, ανησυχίε. Τα μεγαλύτερα ποσοστά τα βρίσκουμε στους νέους τα υψηλότερα ποσοστά ενεργείας επίσης εντοπίζονται στην Χευρώνα και την Καλκίλια ε, περιοχές που βρίσκονται σε κατάσταση πολιορκίας. Σε μικρότερες κοινότητες όπως η Μπίτου και η Μπάρτα τα ποσοστά ενεργείας έχουν αυξηθεί πάνω από 50% ε, και τα μικρά χωριά των προσφύγων που είχαν καλή οικονομική κατάσταση τώρα απλώς εξαρτώνται από την ανθρωπιστική βοήθεια για τρόφιμα και εμβάσματα για τι οικογένειε καθώ και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να επιβιώσουν. Έτσι λοιπόν υπάρχει και η επισητιστική ανασφάλεια στην Δυτική Όχθη. Μια κοινή μελέτη από την UNRWA, την UNICEF και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων ε, δείχνει ότι το πρόβλημα στην περιοχή είναι οξύτατο. Ε, υπάρχει ένα ποσοστό 79% του πληθυσμού που δεν έχει καμία επισητιστική ασφάλεια, 93% είναι χρεωμένοι, 20% δεν έχουν καμία περαιτέρω ε, πρόσβαση σε πιστώσει. Επίση υπάρχουν ε, σοβαρά προβλήματα στην ε, κατάσταση υγεία. 28,5% των παιδιών ...28% των παιδιών που ε, βρίσκονται σε κατάσταση υποσυτισμού, 15,3% κάτω από το κανονικό βάρο, 5,9% ε, έχουν ε, διαρκή οξία έλλειψη τροφίμων. Εδώ λοιπόν δεν φαίνονται να υπάρχουν τίποτε σημάδια βελτίωση, ιδίως ε, στη Δυτική Όχθη αλλά και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Υπάρχουν ε, περιοχές της πόλης που ελέγχονται ακόμη πιο αυστηρά και βρίσκονται στα κατάσταση πολιορκίας ε, σε σχέση με την υπόλοιπη Παλαιστίνη. Στην Ανατολική Ιερουσαλήμ ουσιαστικά έχουμε μια κατάσταση των προαστίων που είναι φτιαγμένα από τενεκεδουπόλεις, μας λένε οι θύνοντες του Γιούνρα. Και αυτό είναι κάτι που έχει ξεκινήσει τα τελευταία δέκα χρόνια και ολοένα και επιταχύνεται ω φαινόμενο. Τώρα, η βία και τα φαινόμενα και η κατάσταση ανασφάλεια για την καθημερινή ζωή των προσφύγων στη Δυτική Όχθη συνεχώ αυξάνονται. Υπάρχουν προβλήματα με τι ένοπλε συγκρούσει και οι κατοικοί στι πέντε μεγαλύτερε περιοχέ όπου δρούν ε, οι ένοπλε δυνάμει ε, βρίσκονται σε κατάσταση πραγματικού κινδύνου. Το κλίμα βεβαιότητα ε, στο πολιτικό επίπεδο λόγω της κατάστασης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, της δυνατότητας εσωτερικής ε, συμφιλίωσης των Παλαιστινίων, ε, η μελλοντική ηγεσία της Παλαιστινικής, αρχή, Αρχής, το τι θα γίνει με τις μελλοντικές εκλογές, όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν το κοινωνικό περιβάλλον και το περιβάλλον ασφαλείας καθώς και τις οικονομικές προοπτικές της περιοχής. Επειδή δεν υπάρχει σαφήνεια για τα θέματα αυτά, οι κάτοικοι γίνονται, είναι συνεχώς σε κατάσταση άγχους, καχυποψίας, και συναισθηματικά δεν μπορούν να ξέρουν ποιε είναι οι ελπίδε του ε, και οι προοπτικέ του για μια καλύτερη ζωή. Η κατάσταση λοιπόν ε, κατοχής ε, και πολιορχίας καθώς και δυνατο... η αδυναμία να έχει κάνει πρόσβαση στην καλλιεργήσιμη γη και την θάλασσα, το 60% δηλαδή τη ε, δυτική όχθη. αυτό υπονομεύει την κοινωνική και οικονομική προοπτική ανάπτυξης της δυτικής όχθης. Κυρίε και κύριοι, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σα. Χρειάζεται να έχουμε θετικές προσπάθειες ανάπτυξης ε, στην πράξη και όχι μικρέ ε, κινήσει. Ε, εδώ πρέπει να αρθεί το καθεστώς ελέγχου, να υπάρξει μια πραγματική επέκταση του χώρου και της ενδυνάμωσης του λαού των Παλαιστινίων για να μπορέσουν οι ίδιοι να, να πάρουν στα χέρια τους την ανάπτυξη ενός, ε, μιας βιώσιμης περιοχής ειρήνης. Επίσης να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, μια περιοχή όπου θέλουμε να διασφαλίσουμε κοινωνική ειρήνη και οικονομική ανάπτυξη. Εδώ τα θετικά αποτελε... Ε, επιτεύγματα της Παλαιστινικής Αρχής μας επιτρέπουν να έχουμε ελπίδες για μια ευημερούσα χώρα που να βασίζεται στην ειρήνη για να ζήσει αρμονικά με τους γειτονές της. Ε, στηριζόμαστε και στις πολιτικές σας πρωτοβουλίες για να ενισχύσουμε την ειρήνη στην περιοχή και αυτό είναι το κλειδί για τα πάντα, αρχή και το τέλος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας ερευνητικού και ενημερωτικού κέντρου Ισραήλ Παλαιστίνης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κυρία Κρέτου. Εκλήθηκα σήμερα στην ακρόαση αυτή για να εκπροσωπήσω ως ε, μέλος του Γητικού Συμβουλίου το IPRC. Είμαι και μέλος ε, του κοινοβουλίου μου, μέρος του ΠΙΕΛΟ και διερωτώ με γιατί εστάλησε εμένα η πρόσκληση, ίσως διότι έχει να κάνει ακρόαση με την οικονομική ανάπτυξη. Εκπροσωπώ επίσης τους Παλαιστινίους ως πρόεδρος του Οικονομικού Κοινωνικού Συμβουλίου της Παλαιστίνης και συγχρόνως είμαι πρόεδρος του Ευρωπαλαιστινιακού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Ως πρόσωπος όμως αυτού του ερευνητικού και ενημερωτικού κέντρου του Ισραηλινο-Παλαιστινιακού, αρχίζοντας θα πω το εξής. Εμείς οι Παλαιστίνοι προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τους γείτονες μας Ισραηλινούς Ισραηλούς σε όλους τους τομείς, τον οικονομικό, τον πολιτικό, διότι θέλουμε να σταματήσει η κατοχή θέλουμε να φτάσουμε στην ε, προσφυλή λύση των δύο κρατών και να έχουμε ένα ανεξάρτητο Παλαιστινικό κράτος δίπλα στο Ισραήλ. Από οικονομικής πλευράς και δεδομένου ότι σήμερα αυτό είναι το θέμα που μας απασχολεί και είμαι ευγνώμων στους συναδέλφους της UNRWA που εξέφρασαν την ε, ανθρωπιστικό ε, πρόβλημα που υπάρχει στη Λωρή της Γάζας και στη Δυτική Οχθή θα πω το εξή. Εμείς εργαζόμαστε για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την οικονομία της Παλαιστίνης και πρόκειται για ένα θέμα πολύ σημαντικό για μας διότι θέλουμε να είμαστε αυτάρκεις, να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις φυσικές μας ανάγκες και στις αναπτυξιακές μας ανάγκες, αλλά ζούμε σε κάτω από πολύ δύσκολες περιοριστικές συνθήκες. Έφεραν οι συνάδελφοι το όλο θέμα, σας είπαν τι σημαίνει στη Δυτική Όχθη, τι συμβαίνει στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά παρόλα αυτά ο κύριος, με τον κύριο Σίμχα στο Τελαβίβ θεσπίσαμε το ε, φόρουμ επιχειρηματιών Ισραήλ-Παλαιστίνης για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ομαλές σχέσεις και να ξεπεράσουμε κάποια από τα εμπόδια. Όπως γνωρίζουν όλοι πάρα πολύ καλά, έχουμε περίπου 660 σημεία ελέγχου που παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία. Το μεγαλύτερό μας πρόβλημα είναι η πρόσβαση και η κίνηση, η μετακίνηση. Εμείς προσπαθούμε το θέμα αυτό να το επιλύσουμε με τους Ισραηλινούς. Είχαμε πρόσφατα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης μία συνάντηση με τον υπεύθυνο δηλαδή της οικονομικής ανάπτυξης και των διεθνών σχέσεων, τον Υπουργό Σιλβάν Σαρόν και καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι και θέσαμε τρία βασικά θέματα. Πρώτα απ' όλα, πρόσβαση και μετακίνηση. Είπαμε ότι μιλάει για οικονομική ειρήνη ο Πρωθυπουργός σας δεν είμαστε κατά της οικονομικής ειρήνης, αλλά θέλουμε πραγματικά να υπάρχει σοβαρή διαδικασία ανάπτυξης της οικονομίας Παλαιστίνης. Ο Πρωθυπουργός Σαλάμ Φαγιάντ πριν από έξι μήνες παρουσίασε το σχέδιο για τις οικονομικές ε, τα οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικής φύσεως υποδομής για να ενισχύσουμε τα θεσμικά μας όργανα σε πνεύμα θετικό. Σε λιγότερο από ένα χρόνο μπόρεσε να θέσει εφαρμογή περίπου 1.500 πρακτικά προγράμματα και σχέδια. Δυστυχώς τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται στην περιοχή Α και Β και όχι στην περιοχή Γ. Αναφέρθηκε εδώ ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδα της Γάδας βρίσκεται υπό την ηγεσία των στρατιωτικών αρχών του Ισραήλ. Περιοχή Γ. Οι περιοχές Α και Β κατά 40%. Επίσης, στην ε, περιοχή Β ε, κανονικά θα έπρεπε όλα αυτά να τα μοιραζόμαστε από κοινού με το Ισραήλ. Είναι καλύτερα τα πράγματα στην ε, περιοχή Α και Β. Στην περιοχή Γ δεν έχουμε καθόλου την κατάσταση. Όλα είναι υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ και της IDF, της Διεθνούς Αυτής Δύναμης και θα μπορούσαμε να μιλάμε για στρατιωτική διοίκηση μάλλον στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πρέπει να έχουμε άδειες για οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε στην περιοχή γάμα της ε, Λωρίδας της Γάζας και είπαμε στον κύριο Σαλόμ για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την οικονομία μας και να μπορέσουμε να είμαστε αυτάρκης και ανεξάρτητοι θα πρέπει να μπορέσουμε όλα τα, τα και τα μπλόκα που υπάρχουν στις, ε, στις διάφορες αρτηρίες να μπορέσουμε να τα άρουμε. Υπάρχουν περισσότερα από 30 και για να μπορέσουμε να κάνουμε business θα πρέπει να μπορούμε να ελέγχουμε τα σύνορα. Πράγμα που όπως γνωρίζετε δεν συμβαίνει. Τα σύνορά μας προς την ε, Αίγυπτο είναι πιο μακριά. Αλλά τα κοντινά μας τα σύνορα είναι υπό τον πλήρη έλεγχο των αρχών του Ισραήλ. Οι εξαγωγές μας δεν μπορούν να βγουν από τη χώρα. Και αν θέλει κάποιος να αναπτύξει οικονομική δραστηριότητα, πρέπει να μπορεί ελεύθερα να εξάγει τα προϊόντα που παράγει. Όλες οι εξαγωγές ε, τη Παλαιστίνη περνάνε από έλεγχο ασφαλεία. Το ίδιο και οι εισαγωγέ προϊόντων. Εάν λοιπόν δεν αρθούν αυτά τα εμπόδια, και θα σας πω γιατί πρέπει να αρθούν με αυτό το παράδειγμα, στην Παλαιστίνη έχουμε μία από τις καλύτερες φαρμακοβιομηχανίες στην περιοχή της Ραμάλα. Και μπορέσαμε στις αραβικές χώρες μέχρι τώρα να εξάγουμε φαρμακευτικά προϊόντα, ακόμη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε πρόβλημα για να εξάγουμε τα προϊόντα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να το κάνουμε πρέπει τα προϊόντα μας από το εργοστάσιο της Ραμάλα να πάνε στους ε, λιανοπολιτές ε, στην Ευρώπη, στη Γερμανία συγκεκριμένα, χωρί να ανοίξουν οι συσκευασίε. Μιλάμε για φαρμακευτικά προϊόντα, για φάρμακα. Και με του περιορισμού που μας θέτει το Ισραήλ, αυτά τα προϊόντα ανοίγονται από τους Ισραηλινούς. Όλα τα φορτία φτάνουν με ανοιχτά τα φάρμακα. Διότι τα ανοίγουν, τα ελέγχουν και μετά θέλουν να τα ξανακλίνουν, τα ξανασφραγίζουν και τα στέλνουν. Κάτι τέτοιο όμω δεν είναι δυνατόν να γίνεται. Οι επιχειρηματίε μα θέλουν να κάνουν business, να αρχίσουν επιχειρηματικέ δραστηριότητε. Στην... Επίση υπάρχει μια κοινή επιχείρηση στην οποία θα θέλαμε να μπορούμε να βοηθήσουμε για να μπορούμε να εξάγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ε, αφαιθούμε μόνοι μας δεν θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε τίποτε. Δεν καν τον τουρισμό μας, πόσο μάλλον τις εξαγωγές μας. Στα θέματα τα τουριστικά επίσης συνεργαζόμαστε με το Ισραήλ, διότι ο τουρισμός είναι ένα από τους πιο σημαντικούς παράγοντες εξέλιξης για το μέλλον και ένας εξαιρετικός τρόπος για να φτάνουν ξένα νομίσματα στο Παλαιστίνη. Και ακόμη είναι πάρα πολύ δύσκολο για την ε, υπουργό τουρισμού μας που ζει στη Βιθλέμ που έχει ήδη συνεργαστεί με τους υπουργούς τουρισμού του Ισραήλ σήμερα να εργαστεί με τον σημερινό υπουργό τουρισμού που εκπροσωπεί τον κύριο Λίμπερμαν από το Ισραήλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν την κατάσταση αγαπητοί συνάδελφοι. Κανένας δεν μπορεί να δουλέψει τον κύριο Άβιγκτορ Λίμπερμαν Είπαμε λοιπόν αυτά τα πράγματα στον κύριο Σιλβά Σαλόν και πιστεύω ότι αυτό που χρειαζόμαστε και αυτό επιμείναμε και το είπαμε και στον κύριο Σαρόν. εάν το σχέδιο ανάπτυξης Παλαιστίνης του δόκτωρα Φαγιάντ και τα σχέδια οικονομικής ειρήνης του κυρίου Νετανιάχου μπορούν να δουλέψουν, θα πρέπει οι Ισραηλινές αρχές να επιστρέψουν στους επιχειρηματίους Παλαιστινίους να αναπτύξουν δραστηριότητες στην περιοχή Γάμα, ΣΥ, διότι εκεί είναι η μόνη δυνατότητα που έχουμε να αναπτυχθούμε. Τώρα δεν θα σας μιλήσω για το τείχος, δεν θα σας... γιατί εδώ μιλάμε για ανάπτυξη, δεν θα σας μιλήσω για κατάσχεση γεών ο μόνος τομέας που μπορούν να εκμεταλλευτούν ακόμη και να συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται επιχειρηματίες και να αναπτύσσονται είναι η περιοχή C, περιοχή Γ. Αν λοιπόν δεν γίνει κάτι τέτοιο, μόνο για διεθνείς σχέσεις, ε, για δημόσιες σχέσεις θα μιλά όταν μιλάει ο Νετανιάχου για οικονομική ανάπτυξη και για οικονομική ειρήνη. Επιτρέψτε μου τώρα να αναφέρω το θέμα το που μας απασχολεί πιο πολύ απ' όλα. Τη λωρίδα της Γάζας. Ο... Με... Τον κύριο Σιλβάν Σαλόμ. Θέλετε να τιμωρήσετε τη Χαμάς το που κάνετε είναι συλλογική τιμωρία όλου του 1,5 εκατομμυρίου Παλαιστινίων που ζει στη λωρίδα της Γάζας. Δεν τιμωρείτε τη Χαμάς, αλλά τους ανθρώπους. Και έτσι έχουμε στην περιοχή αυτή ανεργία πάνω από 50%, 80% των οικογενειών στη λωρίδα της Γάζας ζουν κάτω από το επίπεδο της φτώχειας και πολλά δεινά ακόμη. Στην περιοχή της Γάζα υπάρχουν ακόμη σημαντικές εγκαταστάσεις και εργοστάσια που πρέπει να έχουν άδεια για να εισάγουν πρώτες ύλες για να ε, δουλέψουν. Με το εμπάργκο δεν γίνεται τίποτα. Απέλησαν το προσωπικό, έκλεισαν τα εργοστάσια. Και έτσι βρίσκονται σε δινή κατάσταση οι κάτοικοι της περιοχής. Για να αναπτυχθεί η οικονομία της περιοχής θα πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Η σύραγγα, οι σύραγγες μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου είναι σημαντική πηγή εσόδων για την Χαμάς. εάν δεν αποκατασταθεί η κατάσταση ε, στη λωρίδα της Γάζα, τα πράγματα θα δυσκολέψουν πολύ περισσότερο. Πρέπει να ξέρετε ότι περισσότερο από το ίμιση του ε, προϋπολογισμού της Παλαιστίνης, της Παλαιστινικής Αρχής στη Ραμάλα, 120 εκατομμύρια δολάρια μηνιαίως υποστηρίζουν τις ανθρωπιστικές ανάγκες και πληρώνουν τις αμοιβέ των δημοσίων υπαλλήλων στη Λωρίδα της Γάζας. 1,5 δις βοήθεια πηγαίνει για τη βοήθεια των Παλαιστινίων της Λωρίδας της Γάζας. Ο δόκτωρ Σαγέντ για φέτος ανήγγειλε ότι θα μπορέσουμε από τον προϋπολογισμό να βοηθήσουμε την περιοχή αυτή με ποσοστό 10%. Πέρσι είχαμε ε, όλο το ποσό που μπορέσαμε να διαθέσουμε για την υποστήριξη της Λωρίδας της Γάζας. Φέτος μόνο 1,2 δις θα χορηγήσουμε για τη Λωρίδα της Γάζας και 300 εκατομμύρια επίσης από την, ε, για την ε, Παλαιστινιακή Αρχή. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την περιοχή μα. Πέρσι η ανάπτυξη όχθητα τη ήταν 6-7%. Ελπίζουμε και φέτο να έχουμε τέτοιου είδου καλά ποσοστά, αλλά αυτό το οποίο πρέπει πραγματικά να μπορέσουμε να κάνουμε είναι να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε όλα τα έργα υποδομή σε όλη την περιοχή. Τώρα, θα σα μιλήσω για την Ιερουσαλήμ, στην οποία γεννήθηκα και μεγάλωσα. Θα τελειώσω σε δύο λεπτά. Η Ιερουσαλήμ περιτριγυρίζεται από οικισμούς Ισραηλινών. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω, διότι έχει περιχαρακωθεί. Τώρα, αυτό το γεγονός αρχίζει και επεκτάνεται και σε εσωτερικές συνοικίες της πόλης της Ιερουσαλήμ. Οι Παλαιστίνοι που ζουν στην περιοχή Ζάχα εκδιώχθησαν διότι κάποιος είπε ότι τα σπίτια τους ανήκαν στην, ε, στο Ισραήλ. Εγώ έχω γεννηθεί στη Ιερουσαλήμ, κοντά στο δρόμο για την Χευρώνα και δεν είμαι ο μόνος, αλλά πολλοί από εμά δεν μπορούν να ξαναγυρίσουν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, στην οποία κατοικούσαν. Πρόκειται λοιπόν για προβοκάτσια. Και έτσι η ειρηνευτική διαδικασία που έπρεπε να αρχίσει πρόσφατα έχει κολλήσει και δεν γίνεται κανένα βήμα προς τα μπρος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για τις παρουσιάσεις σας. Τώρα έχουμε λιγότερο από μισή ώρα για να κάνουμε ερωτήσεις και να ακούσουμε τις απαντήσεις σας. Ο κάθε συνάδελφος να λέει μέλος ποιας Επιτροπής είναι η ποια αντιπροσωπείας και σε ποιον απευθύνει την ερώτησή του. Τρεις ερωτήσεις κάθε φορά. Η κυρία Μπερνά, την πρώτη ερώτηση. Είμαι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Κοινοβουλευτικής ε, Συνέλευσης για την ε, Ευρώπη και το Μεσόγειο. Ήθελα να πω ότι η ειρηνευτική διαδικασία πρέπει να είναι, καθεστώ, να είναι μια διαδικασία ε, παύση του επικισμού. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια συνεχή πολιτική, διαρκή πολιτική επικισμού, που ουσιαστικά είναι η τακτική πολιτική Νατανιάχου, Λίμπερμαν και του σιωνιστικού ε, κράτους. Είναι ίσως ένα εργαλείο, ένα μέσο για να καταπολεμάται η ειρήνη, αλλά για να την πετύχουμε την ειρήνη πρέπει να σταματήσει όλη αυτή η πολιτική. Να θυμίσω εδώ μια απόφαση του ΔΕΚ 26 Φεβρουαρίου, της 26 Φεβρουαρίου που καταλήγει ότι οι τελωνιακέ υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκής Ένωση δεν μπορούν να δίνουν πρωτομησιακό καθεστώ στα προϊόντα τη ε, της εάν έρχονται με πιστοποιητικά του Ισραήλ. Πρέπει να πω ότι στην περιοχή συνάντησα κάποιους συνομιλητές, ε, μεταξύ των οποίων και εκπροσώπους του οργανισμού Γιούντα, και εδώ χαιρετίζω και το έργο που κάνετε εκεί, αλλά να πω δύο πράγματα. Ότι τα προϊόντα που είναι συνήθως γεωργικά, όπως οι φράουλες που παράγονται στην γλώσσα της Γάζας ουσιαστικά με μέσα απατηλά ε, τελικά έχουν ετικέτες ψευδείς, οι οποίες αναφέρουν ότι είναι Ισραηλινής προέλευσης. Είναι λοιπόν ε, παραπημένες οι ετικέτες τα προϊόντα αυτά. Και έχω και μια δεύτερη παρατήρηση, ερώτηση. Εντάξει, μία και μόνη. Ωραία. Ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, Θα συνεχίσω στα ρωμανικά. Είμαι μέλος της Επιτροπής IPRE και μέλος της αποστολής ε, για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη. Πρόκειται για μια στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και προφανώς θα πρέπει να συμμετάσχει πιο πολύ στην διαδικασία αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια πολύ σημαντική πτυχή στη συνεργασία μεταξύ Ένωσης και Παλαιστινιακής Αρχής είναι η οικονομική πτυχή και η ανθρωπιστική βοήθεια. Να σας υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί το βασικό εταίρο Συρίας, Λιβάνου, Αιγύπτου, Σαουδικής Αραβίας, όχι μόνο του Ισραήλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί και τον βασικό δωρητή προς ε, την Παλαιστινιακή Αρχή με συνεισφορά πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ. Επίσης, ε, συμμετέχουμε και μέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Είναι σημαντικό λοιπόν θεωρώ να σας υπενθυμίσω σε όλους ότι η οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να επικεντρωθεί στην, και να συνεχίσει να επικεντρώνεται στην περιοχή αυτή παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα τερμαστεί ο πόλεμος. Είμαι βέβαιος ότι οι δραστηριότητες θα στεφτούν με επιτυχία αλλά όσο ένας από τους δύο εταίρους διέρχεται οικονομική κρίση, θεωρείται ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική ανάκαμψη της περιοχής υπό την Παλαιστινιακή Αρχή αποτελεί βασικό παράγοντα για τον τερματισμό των εχθροπρακτιών. Σας ευχαριστώ. Αξιότιμα μέλη του πάνελ, θα μιλήσω στα σλοβενικά. Να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε για να συζητήσουμε μια πολύ σημαντική πτυχή της ε, σύγκρουσης Παλαιστίνης και Ισραήλ και εννοώ την πτυχή της οικοδόμησης ε, γεφυρών για την οικονομική πρόοδο και ανάκαμψη. Νομίζω ότι πρόκειται για μία μοναδική και πάρα πολύ κρίσιμη ευκαιρία. Κατά κάποιο τρόπο δοκιμάζομαι για το κατά πόσο μπορούμε να ανοίξουμε και μία άλλη διάσταση σε αυτή την σύγκρουση. Φυσικά κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στον ίδιο τον εαυτό και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπε η κυρία Σινιώρα, ότι ουσιαστικά οτιδήποτε συζητάμε, είτε η πτυχή της οικονομίας, είτε η πτυχή της ασφάλειας, η κατάσταση των κατεχομένων, όλα αυτά έχουν νόημα μόνο αν ενταχθούν στο πλαίσιο δύο κυρίαρχων κρατών, τα οποία θα πρέπει να εξέλθουν από την κατάσταση αυτή, να αναγνωρίσουν το ένα το άλλο, να συνεπάρξουν ειρηνικά προκειμένου να εγγυηθούν το ένα στο άλλο την ειρήνη και την ασφάλεια. Οτιδήποτε δεν εντάσσεται στο πλαίσιο αυτό είναι δευτερευούση σημασία, αν θέλετε. Θεωρώ ότι έχουμε επαρκείς λόγους και ακούσαμε κάποια από τα επιχειρήματα σήμερα για να έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι να αμφισβητήσουμε το ότι βελτιώνεται η κατάσταση επί τόπου και το Ισραήλ σκοπεύει να συνεχίσει στο ρόλο του κράτους μέλους που κατέχει και περιορίζει την ελευθερία της κυκλοφορίας, για παράδειγμα. Όλα αυτά αποτελούν απαραίτητους όρους για μια φυσιολογική οικονομική ανάπτυξη. Αυτή η πολιτική κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχιστεί. Θα σταματήσω στο σημείο αυτό γιατί δεν έχει νόημα να συζητάμε σε αυτό το πλαίσιο. Καλωσορίζω την καλή θέληση που υπάρχει από αμφότερες τις πλευρές και από τους εκπροσώπους και της Παλαιστινιακής και της Ισραηλινής πλευράς εδώ. Αλλά η ερώτησή μου εν τέλει θα θέσω Μία ερώτηση μόνο, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα που θα παραμείνουν ανοιχτά. Να μου πείτε τι γίνεται με την προσβασιμότητα στην ανθρωπιστική βοήθεια. Γιατί έχω επισκεφθεί κάποιες φορές τη Μέση Ανατολή και κάθε φορά μου λένε ότι οι Ισραηλινές αρχές εκμεταλλεύονται τον έλεγχο που ασκούν για να περιορίσουν την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια. Δηλαδή ότι επινοούν διάφορα γραφειοκρατικά εμπόδια, αλλάζουν τους καταλόγους των ε, προϊόντων που μπορεί να χορηγηθούν μέσα σε μία νύχτα, προκειμένου να δυσκολέψουν το έργο της ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτό αληθεύει και θα ήθελα να ακούσω μία απάντηση από αυτούς που ασχολούνται καθημερινά με τέτοια θέματα. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Δεν ξέρω ποιος από τους ομιλητές μας θα θέλει να πάρει το λόγο για να απαντήσει. Δεν υπήρξε κάποια ερώτηση συγκεκριμένα προς κάποιον από το πάνελ μας. Εκτός μικροφώνου σχόλια. Ε, Για τη λωρίδα της Γάζας. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι όπως έχουν η κατάσταση, όπως έχει η κατάσταση σήμερα, η ανάπτυξη είναι πάρα πολύ δύσκολα. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, καταβάλουμε κάθε προσπάθεια. Ωστόσο, υπό τις παρούσες συνθήκες έλλειψης πρόσβασης, έλλειψης ελευθερίας κυκλοφορίας και όσο συμβαίνει στη λωρίδα της Γάζας, είναι πολύ δύσκολο να διανοηθούμε ότι θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την οικονομική μας υποδομή. Αν μου επιτρέπετε, και αυτό μας το είπαν και στη Γάζα, ε, η Γάζα θέλει να ανακάμψει σαν την Ανδώρα. Δεν μπορεί να κατασκευάσει. Θέλει να αποτελέσει εμπορικό κόμβο. Γιατί εμπορικό κόμβο αποτελούσε και με τους Αιγύπτιους. Τότε με τον Άσαρ όλοι οι Αιγύπτιοι πήγαν για ψώνια στην ε, Γάζα. Και νομίζω ότι αυτό το παράδειγμα μπορεί να συνεχιστεί στο μέλλον αλλά αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα γιατί δεν έχουμε ειρήνη. Αν τραυματιστεί η κατοχή, αν επικρατήσει η ειρήνη, νομίζω ότι οι κάτοικοι της Γάζα όχι μόνο θα καλωσορίσουν και τους Αιγυπτίους και τους Παλαιστινίους και του καθεξής, αλλά θα θέλουν και εμπορικές σχέσεις με τους Ισραηλινούς. Γιατί και οι Ισραηλινοί ερχόντουσαν στη λόγια της Γάζας, όταν τα πράγματα ήταν καλύτερα. Αν θέλετε να προσθέσετε κι εσείς κάτι. Ναι, αναφέρατε την ε, πρόσβαση στη βοήθεια. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, ιδιαίτερα για τη Γάζα. και τα πράγματα είναι περιορισμένα και στην δυτική όχθη. Είναι δύσκολο κανεί να έχει πρόσβαση στην διοικητική όχθη. Υπάρχουν διοικητικοί περιορισμοί, είναι πάρα πολύ δύσκολοι και για το προσωπικό να μετακινηθεί στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Υπάρχουν σημεία ελέγχου. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Και νομίζω ότι και η κυβέρνηση του Ισραήλ κατανοεί ότι το έργο μας και το έργο των άλλων οργανώσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι θα μπορούσαν να κάνουν πιο πολλά για να διευκολύνουν το έργο μας και προσπαθούμε να επιστήσουμε την προσοχή τους ε, στα εμπόδια αυτά. Γιατί Γάζα τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Μάξ, δεν ξέρω αν θέλεις να πάρεις το λόγο. Uh, πολύ σύντομα για τη Γάζα και όπως είπε και η Μπάρμπαρα, πέραν από ένα περιορισμένο αριθμό τροφίμων και άλλων προϊόντων για την ανακόφιση των προσφύγων και κάποιο μετρητό, κάποια από αυτά φτάνουν. Αλλά μιλάμε για μια γκάμα 25-30 προϊόντων. Και κάποτε είχαμε 5-6 χιλιάδες ε, προϊόντα, είδη προϊόντων που διακινούνταν στη Γάζα. Ένα απλό παράδειγμα. Το, η ράβδη τσιμέντου και, και τσαλιού για, να, την ανοικοδόμηση στη Γάζα δεν επιτρέπεται να μπουν. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τις ακούσουμε όλες, αλλά θα κάνουμε και ένα μικρό διάλειμμα πριν το δεύτερο γύρο του, της συζήτησης. Ο κύριος Γκέρενς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σπάνια έχουμε δει τέτοιου κατάσταση. Πήγα από αυτή που είδα στη, Γάζα εδώ και κάποια χρόνια και αυτή τη στιγμή κάποιος λέει ότι τα πράγματα επιδεινώνονται και διαρωτώ τι μπορεί δεδομένης κατάστασης να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο. Πολύ απλή ερώτησή μου. Ήδη αναφέρθηκε ε, αν αναφέρθηκε ένας αριθμός πριν να έρθω, ξεχάσει την ερώτησή μου. Η ερώτησή μου αφορά το σύνολο ε, του ποσού τα οποία από το εξωτερικό μέσο του Ισραήλ πηγαίνουν στο Ισραήλ στην ε, ε, Παλαιστινιακή, Αρχή και για την Δυτική Όχθη και για την Λωρίζα της Γάζας. Παρακαλώ να είστε σύντομοι γιατί έχουμε λιγότερο από 10 λεπτά για τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Ο κύριος Βένσον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνούμε απολύτως ότι όλοι με το ότι θα μπορέσουν να συνεπάρξουν ε, συνειρηνικά αυτές οι δύο χώρες. Θα ήθελα να κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Ξέρουμε ότι το Χαμάς θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση. Και όταν μιλούμε για οικονομική ανάπτυξη, πρέπει να λάβουμε υπόψη την ε, Φατά και την Χαμάς και πρέπει να δούμε τι ακριβώς πηγαίνει, τι συμβαίνει στην περιοχή και κυρίως ποια είναι η θέση του Χαμάς στη λωρίδα της Γάζα. Ξέρουμε ότι η λωρίδα της ε, Γάζα ήταν μια οικονομικά εύρωστη περιοχή και ήταν πάρα πολύ η σημαντική για τις συναλλαγές με την ε, Γάζα. το ότι η Γάζα κυβερνάται από το Χαμάς τι σημαίνει για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και ποιος είναι ο ρόλος που στην πραγματικότητα παίζει για την περιοχή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συμμετείχα σε μια διεθνή συνάντηση την Πέμπτη σε ό,τι αφορά τα θέματα των φίλων για την Μέση Ανατολή και συμμετείχαν και εκπρόσωποι του Κουαρτέτου αλλά και εκπρόσωποι, γυναίκες εκπρόσωποι από την Παλαιστίνη και το Ισραήλ και εξέφρασαν το εξής ότι απομακρυνόμαστε από μια λύση δύο κρατών και ότι ο πληθυσμός ε, στην Παλαιστίνη έχει κουραστεί και δεν διαβλέπει πλέον να υπάρχουν πρόπτικες. Δεν υπάρχει πλέον να ε, φαίνεται προθυμία της κοινωνίας των πολιτών να μειχθεί στο θέμα αυτό. Μιλήσατε για την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στην Δυτική Όχθη και στη Γάζα και παρευρέθηκα στη Γάζα τον Ιανουάριο, τα είδα πράγματα με τα ίδια μου τα μάτια. Η πολιτική θέληση εξακολουθεί να λείπει για την εξέβρεση λύσης από όλες τις πλευρές. Γι' αυτό να σας ρωτήσω κυρία Σενιόρε και και εσάς κύριε Σίμχα, το εξής. Ποια πολιτικά βήματα θεωρείτε ότι είναι ρεαλιστικά στην παρούσα κατάσταση και στο Ισραήλ αλλά και στην Παλαιστίνη προκειμένου να εξέλθουμε από το διέξοδο αυτό. Μπορεί να γίνει κάτι με την διεθνή διαμεσολάβηση. Ποια είναι, ποιος είναι ο πολιτικός ρόλος που πρέπει να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρα από την ανθρωπιστική βοήθεια και ποια βήματα πρέπει να γίνουν από την Παλαιστινιακή Αρχή σε ό,τι αφορά την ε, εσωτερική Παλαιστινιακή κατάσταση και τι μπορεί να κάνει από πλευρά του και το Ισραήλ. Αυτά σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τρεις ερωτήσεις ακόμα, λέει η Πρόεδρος. Ε, thank you very much. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ δεν είπατε. Ωραία. συμμετέχω στην αποστολή στην Παλαιστινιακή Αρχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είμαι και μέλος της ομάδας εργασίας για την Μέση Ανατολή. Επισκέφθηκα την Γάζα και τη Δυτική Όχθη πρόσφατα το Σεπτέμβριο και τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, λίγο μετά την επίθεση στη Γάζα και αυτά που μας λέτε εδώ σήμερα μου καταδεικνύουν ότι πολύ απλά δεν, υπήρχε, δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή σε σχέση με αυτά που είδα πριν από ένα χρόνο και αυτό είναι φρικιαστικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μία από τις πιο ισχυρές πολιτικές ε, και οικονομικές σχέσεις με το Ισραήλ. Ουσιαστικά σε σχέση με καθ' άλλη χώρα εκτός της Ένωσης. Άρα λογικά η σχέση θα έπρεπε να είναι αρκετά δυνατή προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να πείσει το Ισραήλ να ανακουφίσει τουλάχιστον, αν, αν, μη τι άλλο, την κατάσταση στην Γάζα. Και νομίζω ότι οι προσπάθειές μας εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούν και στο μέλλον. Εντάλλως, θεωρώ ότι δεν υπάρχει ελπίδα, δυστυχώς, για ειρήνη στην περιοχή. Χαίρομαι που άκουσα τις παρουσιάσεις σας, αλλά μου άρεσε ιδιαίτερα αυτά που μας είπαν οι εκπρόσωποι των επιχειρηματιών, γιατί συνδεθήκαμε τον Φεβρουάριο του περσινού έτους με τους εκπροσώπους του εμπορικού επιμελητηρίου στη, Γάζο, στη Γάζα, των οποίων ε, οι επιχειρήσεις και βιομηχανίες είχαν καταστραφεί πλήρωναν υπέρογκα ποσά για οι πρώτε ύλε και δεν μπορούσαν καν να συνεχίσουν τις εργασίες τους. Είναι σαφές ότι η Παλαιστινιακή οικονομία δεν μπορεί να ευημερήσει, δεν μπορεί ο κόσμος να ευημερήσει. Χρειάζεται ελευθερία διακίνησης, ελευθερία εξαγωγών-εισαγωγών, ελευθερία άσκησης εμπορίου. Είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε γέφυρε, αλλά αυτό που θέλω να πω ότι πέρα από τις συναντήσεις μου πέρσι, είναι η πρώτη φορά που βλέπω εκπρόσωπους των επιχειρήσεων εδώ και νομίζω ότι θα πρέπει να το επαναλάβουμε αυτό πιο συχνά. Θα ήθελα να σας πω ότι γενικά οι επιχειρηματίες διαδραματίζουν πολύ μεγάλο ρόλο για την αλλαγή των κυβερνητικών πολιτικών και να, σε ό,τι αφορά το άνοιγμα των δυνατοτήτων για την ειρήνευση στην περιοχή. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικός και κρίσιμος ο ρόλος που καλείστε να διαδραματίσετε για την οικοδόμηση καλύτερων σχέσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Έχουμε καθυστερήσει. Προτείνω στους συναδέλφους να θέσουν τα ερωτήματά του στην επόμενη ευκαιρία να δώσω το λόγο στο πάνελ για να απαντήσει. Uh, <clears throat> Εάν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να αφαιρθώ σε δύο ερωτήματα που τέθηκαν. Ο κύριος Σούλτς, αν δεν κάνω λάθος πρώτα απ' όλα. Θα αρχίσω με εσά, λοιπόν. Οι επιχειρηματίες στο Ισραήλ έκαναν πολύ καλές επιχειρήσεις και με τη Δυτική και με την περιοχή της Γάζα. Και καταβάλουμε όλες τις προσπάθειες για να ξαναρχίσουμε και πάλι από την αρχή είπα, ευθύ εξ αρχής δεν είμαστε πολιτικοί. Είμαστε εκεί και προσπαθούμε να ασκήσουμε πιέσεις και να επηρεάσουμε τις κυβερνήσεις μας για να κάτσουν από κοινού δύο τραπέζι και να συζητήσουν. Ο μόνος τρόπος είναι να συζητηθούν τα προβλήματα. Πραγματικά πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε διάβλους εμπιστοσύνης και σεβασμού των μεν προς τους δε. Διότι τελικά οι επιχειρήσεις μπορούν να προσεγγίσουν του ανθρώπου. Είναι πραγματικότητα αυτό, δεν είναι σλόγγα. Και τελικά βλέπουμε ότι πολλοί από την Γάζα τηλεφωνούν στους φίλου από το Ισραήλ και του λένε ελπίζουν θα μπορέσουμε να επαναλάβουμε το πείραμα αυτό. Αυτό είναι προ το καλό όλων και κατανοώ ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη στη Γάζα αυτή τη στιγμή και εμείς πραγματικά περιμένουμε στην άκρη. Περιμένουμε να προσεγγίσουμε τους άλλους και να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και μπορώ να σας πω ότι αυτά τα λέω εκπροσωπώντας επιχειρηματίες της περιοχής. Δεν είμαι πολιτικός. Έχουμε γύρω στα 3 δις ε, δολάρια προπολογισμό για την Παλαιστίνη. Η Χαμάς όμως δεν μπόρεσε να φτάσει στις κάλπες. Εάν μπορούσε να κυβερνήσει και για τη στάση που ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ασκώντα εμπάργκο όπω το Ισραήλ και οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, εναντίον τη Χαμά, ε, οδήγησε στη σημερινή κατάσταση. Το ίδιο έγινε και με την Αλγερία στο παρελθόν. Εκεί είχαμε την αντίστοιχη Παλαιστινιακή Αρχή, την Εφελέν, και ξέραμε ότι δρούσαν ε, επηρεαζόμενοι και από ισλαμικές, ισλαμιστικές παρατάξεις στην Αλγερία. Δεν επιτρεπόταν λοιπόν να κυβερνήσουν στην Αλκυρία οι Ισλαμιστικέ παρατάξει και έγινε εμφύλιο πόλεμο που ακόμη και σήμερα έχει φυσικά τα Ακόμη χάνουν τη ζωή του άνθρωποι. Γιατί δεν αφήνουν τι Ισλαμιστικέ παρατάξει να έρθουν στην εξουσία. Λοιπόν, αν η Χαμά είχε τα ενία τη κυβέρνηση, ίσω να είχαν μετριάσει τι ακραίε θέσει του. Ελπίζουμε ότι πριν η συνάντηση του Αραβικού συνδέσμου στις 28 του Μάρτη συζητήσει για την ερευνητική διαδικασία της οποίας έγινε η Αίγυπτος. Ε, ελπίζουμε ότι πρωτού γίνουν όλα αυτά ίσως υπάρξουν κάποια δείγματα επιτυχίας. Αυτό μπορεί να μας επιτρέψει να προχωρήσουμε. Τι πρέπει να κάνει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζω ότι υπήρξατε γενναιόδοροι ιδίω με τους Παλαιστινίου δίνοντας ό,τι περισσότερο μπορείτε. Όμως αυτό που πραγματικά χρειάζεται ο κόσμος εκεί είναι πολιτική συμμετοχή. Πρόσφατα λήφθησαν αποφάσεις στη Μόσχα από το κουαρτέτο. Εκεί δηλώθηκε ότι σε δύο χρόνια θα αναγνωριστεί έναν εξάρτητο Παλαιστινιακό κράτο. Αυτό πρέπει να επιδιώξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωκοινοβούλιο. Δηλαδή τα ερχόμενα δύο χρόνια και αν δεν πετύχει η ειρηνευτική διαδικασία, τότε πραγματικά να κηρυχθεί ανεξαρτησία, να αναγνωριστεί η ανεξαρτησία του Παλαιστινικού κράτου. Και από όλη την διεθνή κοινότητα να αναγνωριστεί. Και παρά του περιορισμού, παρά τι δυσκολίε. Είναι τόσο δύσκολο να έχουμε συνομιλίε με του Ισραηλινού. Παρ' όλα αυτά το κάνουμε. Ακόμη και με άτομα που είναι τόσο δύσκολο να έχει κανεί μαζί του συνομιλίε, όπω ο κ. Σαρών. Και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την ειρήνη. Πρόεδρο. Ευχαριστούμε πολύ όλου του ομιλητέ μα. Ένα λεπτό διάλειμμα για το δεύτερο πάνελ μα.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 Maybe press will help us Παρακαλώ. Ήρθε η ώρα να αρχίσει η συζήτηση στο δεύτερο πάνελ. So, we came to, πάνελ αυτό οργανώνεται σε συνεργασία με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καλωσορίζω τον κύριο Μποντής. Αναμφίβολα, το μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το δεμινάριο οφείλεται στον επόμενο μιλητή μας, τον πρώην Πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας, τον Μπλερ ο οποίο ήρθε από το Ισραήλ σήμερα το πρωί. Ω ειδικό εκπρόσωπος του κουαρτέτου στη Μέση Ανατολή είναι εξοικειωμένο με τις θέσεις των εμπλεκομένων μερών. Όταν σκέφτηκα να οργανώσω ένα σεμινάριο αυτό, είπα ότι θα πρέπει να έχουμε μία προσέγγιση όσο πιο ουδέτερη πολιτικά γίνεται παρά το γεγονός ότι η επίλυση αυτή της σύγκρουση μόνο μπορεί να είναι απόρρια πολιτικών αποφάσεων. Παρ' όλα αυτά, είναι πολλές φορές οι πολιτικές προσεγγίσεις μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένη κατεύθυνση ή σε αδιέξοδο. Κατά συνέπεια, επικεντρώσαμε την προσοχή μας, τη συζήτηση μας, την ανάπτυξη, την ανθρωπιστική βοήθεια και στην οικονομική συνεργασία με τη Γάζα και Δυτική Όχθη. Θέλουμε να ακούσουμε την άποψη του Τόνι Μπλε, στον οποίο δίδω αμέσω το λόγο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την δυνατότητα να απευθυνθώ σε εσάς σήμερα. Θα αρχίσω κάνοντας μια γενική επισκόπηση της όλης κατάστασης. Αρχίζοντας όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξή τους και την εργασία που καταβάλουν υπέρ των Παλαιστινίων. Όπως ξέρουμε είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρικτές της Παλαιστινικής Αρχής και θα πω πώς τα κονδύλια που καταβάλουμε ωφελούν τους Παλαιστινίους. Όπως προαναφέρατε. Πραγματικά ήρθα απευθείας από την περιοχή αυτή. Χθες είχαμε συζητήσει στην Ιερουσαλήμ με την ηγεσία του Ισραήλ και πριν από μερικές μέρες συζητήσαμε και με την ηγεσία των Παλαιστινίων και με την ηγεσία των Ισραηλινών για να δούμε πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Ξέρουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, πόσο δύσκολα ήταν τις τελευταίες μέρες. Υπάρχουν δύο βασικά θέματα. Το πρώτο είναι πώς θα προχωρήσουμε από εδώ που βρισκόμαστε σε μια τραγική κατάσταση με απώλειες ζώων, νέων Παλαιστινίων, με μεγάλες εντάσεις μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλών τις τελευταίες μέρες, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε πολιτική διαπραγμάτευση και δεύτερον, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η Παλαιστινιακό κράτος θα είναι μία λύση πραγματική για αύριο και πώς οι προσδοκίες των Παλαιστινίων θα μπορέσουν η δημιουργία του κράτους να υλοποιηθεί. Τώρα, όσον αφορά τις πολιτικές διαπραγματεύσεις, όπως ξέρετε, η ιδέα είναι να μπορέσουμε να έχουμε συνομιλίες μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών τις επόμενες μέρες και τις επόμενες εβδομάδες και μήνες να μπορέσουμε να τους κάνουμε να διαπραγματευτούν όλα τα θέματα τα οποία τους απασχολούν. Αύριο ο Πρωθυπουργό του Ισραήλ θα συναντήσει τον Πρόεδρο Ομπάμα στην Ουάσιγκτον. Σε σχέση με την εργασία την οποία εμείς επιτελούμε, εγώ εστιάζομαι στην οικονομία της Παλαιστίνης και την δυνατότητα που, έχουν έχει η Παλαιστινιακή Αρχή να μπορέσει να, να η, η δική μου προσέγγιση είναι, πιστεύω, από κάτω προς την κορυφή της πυραμίδας και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, θέλουμε μία λύση με δύο κράτη. Η μόνη βάση, βάση της οποίας μπορούμε να προχωρήσουμε, είναι μία βάση στην οποία θα είναι σίγουρο το Ισραήλ ότι θα είναι εγγυημένη η ασφάλειά του. Και οι Παλαιστινοί θα πιστεύουν ότι αν θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό, θα μπορέσουν να έχουν ένα κράτος το οποίο να λειτουργεί σωστά. με ένα ξάρτο, κράτος ανεξάρτητο, βιώσιμο, το οποίο να λειτουργεί σωστά. Εάν το κάνουμε αυτό, με την δημιουργία θεσμικών οργάνων, κάνοντας ένα κράτος δικαίου με συνθήκες ασφαλείας, όλα θα είναι κατά. Και αυτό προσπαθούμε να υλοποιήσουμε εσύ. Το 2007 ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία με την υποστήριξη της ε, Γαλλίας που οργάνωσε την διάσκεψη, την ε, αρχική που είδε στον Ακτήριο λάσκτισμα και με την ε, συμβολή των διεθνών δυνάμεων. Και πρέπει να πω ότι τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι έχει γίνει σημαντική πρόοδος στη θεσμικά όργανα του Παλαιστία. Σήμερα στη Δυτική Όχθη, παρά τι δυσκολίε και τα προβλήματα που υπάρχουν, η Παλαιστινιακή Αρχή υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού Φαγιάντα έχει αναλάβει ένα πρόγραμμα δημιουργίας ενός κράτου δικαίου και εκεί βασίζεται και η δική μας υποστήριξη Στις περισσότερες πόλεις και περιοχές της Δυτικής Όχθης η υπεύθυνη για την τάξη και την ασφάλεια είναι η αστυνομία της Παλαιστίνης. Πρέπει να πω ότι με τη συνδρομή των Ευρωπαίων έχουν οι αρχές, οι αστυνομικές και οι δικαστικές ε, ε, βοηθηθεί για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση που δημιουργείται και πιστεύω ότι υπάρχει παρά τις δυσκολίες, αυτή η αυξημένη ικανότητα των Παλαιστινίων να μπορέσουν να χειριστούν αυτά τα θέματα. Τη φορά επίση πρέπει να πω ότι έχει υπάρξει ε, κάποια ε, εν μέρη μικρή μείωση των περιορισμών κυκλοφορίας και πρόσβασης κύριες οδικές αρτηρίες μεταξύ βορρά και νότου, στην δυτική όχθη και πολλά σημεία ελέγχου έχουν ε, ανοίξει, έχουν αρθεί εν μέρη. Η αύξηση της παλαιστινιακής οικονομίας πέρσι ήταν της τάξης του 7% περίπου. Αλλά ακόμη υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Και επιτρέψτε μου να σας κάνω μία μικρή ανάλυση της όλης κατάστασης. Θέλετε να επεκταθώ, να είμαι σύντομα. You want me to go for 50 minutes or you want me less than 50 minutes? do whatever you want. I'm, uh, I'm used to this. Uh, Πόση ώρα έχω στη διάθεσή μου, πείτε μου. Μάλιστα, μην ανησυχείτε θα τελειώσω εντός της προθεσμίας. Αν ε, κοιτάξουμε λοιπόν τα μέτρα επί των οποίων εργαζόμαστε στην παρούσα φάση, καταρχάς προσπαθούμε να πετύχουμε πιο πολύ ασφάλεια και ελευθερία για τις Παλαιστινιακές δυνάμεις. Κατά δεύτερον, τα βασικά βιομηχανικά προγράμματα να ξεκινήσουν στην Δυτική Όχθη. Έχουμε πέντε βιομηχανικά πάρκα τα οποία υποστηρίζουμε, μερικά από τα οποία θα ξεκινήσουν επόμενους μήνες και προγραμματίζονται μεγάλα πακέτα σε ό,τι αφορά τον τουρισμό και άλλα οικονομικά προγράμματα στα Βυτική Όχθη, όλα εκ των οποίων θα βοηθήσουν την ευημερία και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Επίσης, προσπαθούμε να αλλάξει το καθεστώς ε, στο 60% των, ε, της ε, Παλαιστινιακών εδαφών και φυσικά υποστηρίζουμε και το κράτος δικαίου. Ωστόσο, είναι τεράστια τεράστιο το έργο μας σε ό,τι αφορά την Δυτική Όχθη αλλά και τη Γάζα που η κατάσταση παραμένει πολύ κρίσιμα. Σας είπα και προηγουμένως ότι θα πρέπει να αλλάξει η πολιτική σε ό,τι αφορά τη Γάζα. Και όντως τις τελευταίες ημέρες υπήρξε ένα επιπλέον πακέτο, ένα επιπρόσθετο πακέτο ανακούφισης προς τη Γάζα, αλλά η κατάσταση εξακολουθεί να ισχύει ως εξής. Η οικονομία δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως πρέπει όλα περνάνε από υπόγειες ε, οδούς και γι' αυτό λοιπόν υπάρχει ο κίνδυνος να καταλήξουμε σε μια κατάσταση που δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι νόμιμες επιχειρήσεις στη Γάζα και όλα θα λειτουργούν μέσω της μαύρης αγοράς. Άρα προσπαθούμε να αναπτύξουμε έργα υποδομή στη Γάζα αλλά και σε ό,τι αφορά την επανεκκίνηση της οικονομίας. Αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ αν, Ισραηλιν, αν, αν ο Ισραηλινός στρατιώτης ο οποίος κρατιέται θεωρώ ότι αυτό θα ε, βοηθούσε πάρα πολύ την κατάσταση. Για να συνοψίσω λοιπόν πως έχει η κατάσταση. υπάρχουν κάποια βράχη πρόθεσμα θέματα, κατά πόσο μπορούν αυτές οι συζητήσεις να μετατραπούν ε, σε πραγματικές διαπραγματεύσεις. Έχουμε το μακροπρόθεσμο στόχο και ερώτημα των υποδομών σε ό,τι αφορά το κρατός δικαίου και τέτοια θέματα, αλλά και μια ολόκληρη πανοπλία, αν θέλετε, μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο οικοδόμημα θεσμών και κυβερνήσεων, προκειμένου να απομακρυνθούν τα εμπόδια τα οποία πνίγουν την Παλαιστινιακή οικονομία. Και να σας πω και τέλος το εξής, ε, εν είδη εισαγωγής, αν θέλετε. Θεωρώ ότι ως ότου τα περιστατικά μετά το 2000 μάλλον μέχρι το 2000 ε, ήταν ίσως δυνατόν να επιτευχθεί μια συμφωνία ενδεχομένως για τα βασικά ζητήματα σε ό,τι αφορά το τελικό στάτους του Παλαιστινιακού κράτους. Και μετά τη συμφωνία αυτή να προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε την πραγματικότητα σε αυτήν τη συμφωνία. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα μετά την κατάρρευση της ειρηνευτικής διαδικασίας του 2000 βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η πραγματικότητα είναι η εξή. Αν δεν καταφέρουμε να οικοδομήσουμε από τα κάτω προς τα πάνω ένα Παλαιστινιακό κράτος, δεν θα καταφέρουμε να πετύχουμε τίποτε. Πολύ λυπάμαι ότι, πολύ φοβάμαι ότι σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα και γι' αυτό θεωρώ ότι αυτό που κάνει το κουαρτέτο και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ίσονος σημασίας, αλλά βασική σημασίας. Αν μπορέσουμε να οικοδομήσουμε το Παλαιστινιακό κράτο, κράτος από κάτω προς τα πάνω, από τις ρίσεις προς τα πάνω, θα έχουμε πετύχει. Εγώ θεωρώ ότι και οι Παλαιστινία και οι Ισραηλοί θέλουν μια λύση δύο κρατών. Αλλά επίσης ότι πρόκειται για μια κατάσταση κατεπίγουσα, πολύ κρίσιμη και ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου να κάνουμε σημαντικά βήματα προς τα εμπρός. Δεν μπορούμε να αφήσουμε μια πολιτική διαδικασία η οποία είναι νόμιμη και παραγωγική και δεν μπορούμε να αφήσουμε την κατάσταση όσο έχει όχι μόνο στη Δυτική Όχθη αλλά και στη Γάζα. Είναι μοναδικός τρόπος να δώσουμε ελπίδα στον κόσμο εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε να περάσουμε στο δεύτερο γύρο ανταλλαγής απόψεων. Και τώρα το λόγο στην πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξής μας, Εύα Ζολή. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ για να μοιραστείτε μαζί μας τις εμπειρίες σας. Έχετε την εντολή του ειδικού αποσταλμένου του κουαρτέτου εδώ και κάποια χρόνια και ξέρετε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 450 σημεία ελέγχου ενώ μόνον 60 προϊόντα μπορούν να μπουν στο, στην Γάζα παρά το γεγονός ότι ο ΙΕ θεωρεί ότι 9.000 είδη προϊόντων χρειάζονται, είναι αναγκαία Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε πώς σκέφτεστε να διαχειριστείτε το θέμα αυτό, πώς οι έλεγχοι θα πάψουν να αρχίσει το εμπόριο. Δεν γίνεται να υπάρξει ελεύθερη κανονική οικονομική δραστηριότητα με 550, 550 σημεία ελέγχου. Τα 9.000 λοιπόν <clears throat> ήδη που απαιτούνται, <clears throat> πώς θα μπορέσουν να φτάσουν ως τη Γάζα. Και ένα τελευταίο ερώτημα περιμένουμε 60 χρόνια. 60 χρόνια μετά από 40 χρόνια κατοχής. Με συγχωρείτε, κόπηκε το μικρόφωνο μου. Διερωτώμε λοιπόν, τι περιμένουμε τελικά. Ακούμε εδώ ότι έχουν γίνει πολύ λίγα στην πράξη τα τελευταία τρία χρόνια. Ακούσαμε πόσο φρικτή είναι η κατάσταση, ότι υπάρχει συνεχής υποβάθμιση. Γιατί λοιπόν υπάρχουν μονομερείς δηλώσεις από τα δύο κράτη μόνο. Ήθελα την άποψή σας για το θέμα αυτό. First um, Καταρχά, ένα από τα βασικά προβλήματα που έχουμε στο πρόβλημα αυτό είναι ότι όταν λέμε στον κόσμο ότι έχουμε καλέ ειδήσει, όλοι απαντούν με τις κακές ειδήσει, με όλα τα κακά περιστατικά. Και όταν λέμε στον κόσμο τι κακό έχει συμβεί, ουσιαστικά ε, κινδυνεύει κανείς και κινδυνεύει να μην αναφέρει ε, τα θετικά θέματα. Το, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και τα δύο. Μας ρωτήσατε τι έχει επιτευχθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός Εφαγιάντε αξίζει να επενεθεί, γιατί σημείωσε μια πραγματική διαφορά. Πριν από τρία χρόνια όταν ξεκίνησα στη θέση αυτή δεν θα μπορούσα να μεταβώ σε μέρη όπως την Αμπλούς. Στην... Στις περιοχές αυτές έχουν ε, έρθει Άραβες, έχει βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση. Η Παλαιστινιακή Αρχή για πρώτη φορά θα περιορίσει την ενίσχυση σε ένα τρίτο και το δύο τρίτα θα χορηγηθούν από άλλες, από παλαιστινιακές, από παλαιστινιακά εισοδήματα. Και είναι αλήθεια ότι όταν λέτε ότι υπάρχουν 550 σημεία ελέγχου, ότι αυτό θα πρέπει να το αναλύσουμε. Τα βασικά σημεία ελέγχου, τα οποία είναι πολύ πιο περιορισμένα σε αριθμό, εξακολουθούν να υπάρχουν, μερικά εκ των οποίων είναι και ανοιχτά όμως πλέον. Πολλά παραπάνω θα πρέπει να πετύχουμε. Ελπίζουμε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα ανοίξει το βιομηχανικό στο Τζάλιμι και το σχετικό project στη Βιθλεέμ θα ξεκινήσει. Αρχές Ιουνίου θα, θα διοργανωθεί και ένα σχετικό συνέδριο το οποίο ελπίζουμε να έχει καλή συμμετοχή γιατί πέρσι θεώρησε πολλοί κόσμος ότι δεν θα συμμετείχε ο αραβικός κόσμος αλλά παρόλα αυτά ήταν ε, διπλάσεις αριθμό οι συμμετέχοντες. Αυτό φυσικά δεν ε, αναιρεί το γεγονός ότι έχουμε ακόμα μεγάλη απόσταση να καλύψουμε. Άρα να σας πω το εξής. Αν μας το επιστρέψει η πολιτική αν, λέω, εφόσον μας το επιτρέψει η πολιτική, αν μας δώσει το χρόνο και το χώρο, αυτό που κάνει ο Φαγιάντης στην Παλαιστίνη είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, σημαντικό και κρίσιμο. Και να πω ως προς τις μονομερείς ε, δράσεις. Αυτό που έμαθα από την η διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία είναι το εξή. Αυτέ οι δραστηριότητες, οι χειρονομίε, αν θέλετε, είναι πιο σημαντικές για αυτούς που τις πράττουν παρά για αυτούς που τις εισπράττουν, που τις βλέπουν. Το Παλαιστινιακό κράτος θα προκύψει μόνο υπάρξει διαπραγμάτευση. Αυτό που πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε παρόλα αυτά, και θα συμφωνήσω, είναι ότι όπου είναι σαφές και προφανές και αυτό αποτελεί το σαφές μήνυμα μας προς την Παλαιστινιακή Αρχή ότι μπορεί να γίνουν πιο πολλά και μπορώ να σας δώσω πολλά τέτοια παραδείγματα για δράσεις που μπορούν πραγματικά να αναλυφθούν και πολύ πιο γρήγορα γιατί συχνά καθυστερούμε ολόκληρους μήνες για άδεια. Άρα, στο σημείο αυτό να υπάρξει πίεση από Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη ΣΥΠΑ, από το Κουαρτέτο αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά στο τέλος να είμαστε ξεκάθαροι. Η μοναδική λύση η οποία θα διαρκέσει θα είναι μια λύση η οποία θα προκύψει από διαπραγμάτευση. Μάλιστα, ο κύριος Μπούης. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Το κουαρτέτο έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια έμεσων διαπραγματεύσεων εδώ και 10 ημέρε. και ελπίζουμε όλοι ότι θα υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών που θα επιτρέψει την επίτευξη λύση για δύο κράτη. Δυστυχώ η αδιαλαξία τη πολιτική τη κυβέρνηση του Ισραήλ θέτει σε κίνδυνο αυτόν τον στόχο. Το είδαμε μόλι την περασμένη εβδομάδα με την αναγγελία τη δημιουργία 1.600 νέων κατοικιών που είναι παράνομε βάσει του διεθνούς δικαίου στην ε, Λορίδα της Γάζας. Η βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα εμποδίζεται από τα σημεία ελέγχου. Στην Γάζα τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε σχολείο ε, κανονικά. Ε, πολλοί υποφέρουν από υποσυτισμό. Και η μόνη μορφή έκφρασης που έχει απομείνει είναι η βία. Το έγγραφό σας από το Μάιο του 2008 προβλέπει τη δημιουργία ενός Παλαιστινικού κράτους είναι πολύ φιλόδοξο. Όμως τι γίνεται όταν η μία από τις δύο πλευρές δεν σέβεται καθόλου τις διεθνείς της δεσμεύσεις ενώ η άλλη από την άλλη πλευρά δεν καταφέρνει να κάνει τη φωνή της να ακουστεί παρά μόνο με πράξεις βίας. Ήδη από δύο χρόνια είστε ειδικό απεσταλμένος του κουαρτέτου η δική σας θεώρηση για την ε, σύραξη την ε, σύγκρουση αυτή, έχει εξελιχθεί σε αυτά τα δύο χρόνια και τι απολογισμό θα δίνατε για τις δραστηριότητες του κουαρτέτου. Πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε όταν το Ισραήλ, το Ισραήλ συγγνώμη, αναγγέλει την δημιουργία νέων ε, κατοικιών τη στιγμή που έχουν αρχίσει μονομερείς διαπραγματεύσεις και τι μέσα μπορεί κανείς να προβλέψει ώστε να επιχρεώσει το Ισραήλ να σεβαστεί τους νόμους και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τον απολογισμό που αναφέρατε και το ρόλο που έχω να λάβει εγώ, δεν έχω να κάνω με τι πολιτικέ διαπραγματεύσει αυτέ καθεαυτέ, αλλά με την οικοδόμηση των κρατικών θεσμών και των οικονομικών δραστηριοτήτων επιτόπου. Επαναλαμβάνοντα αυτό που μόλι προείπα, νομίζω ότι έχει υπάρξει σοβαρή παρόλα αυτά πρόοδο. Ιδίω με το πρόγραμμα Φαγιάντ που παρουσιάστηκε στη διάσκεψη των Παρισιών του 2007 και την προσπάθεια υλοποίησή του. Νομίζω ότι ρωτήσατε ποια είναι η δική μου θεώρηση και πώς έχει εξελιχθεί την τελευταία διετία. Είμαι ακόμη πιο αποφασισμένος τώρα και θα το λέω με περισσότερη έμφαση ότι ο μόνος τρόπος είναι να υπάρξει μια λύση στον εδαφική στον διαχωρισμό μεταξύ των δύο κρατών. Θα έχετε πάει πολύ ίσως ε, ως εκεί ταξίδι. Ε, μιλάμε για μια μικρή λωρίδα γης. Οι άνθρωποι ζουν ο ένας δίπλα στον άλλον, πάρα πολύ κοντά. Η αλήθεια είναι ότι οι Ισραηλινοί ανησυχούν για την ασφάλεια και από την πλευρά της διεθνούς κοινότητας υπάρχει αρκετή δυσαρέσκεια και θυμός για τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Όντως, όμως υπάρχει πραγματικά πρόβλημα από την πλευρά των Ισραηλινών με την ασφάλεια. Αν αυτό δεν το κατανοήσουμε και δεν το επιλύσουμε, δεν θα καταλάβουμε τις ρίζες του προβλήματος. Ο μόνος τρόπος να επιληθεί το ζήτημα είναι να οικοδομηθούν οι δυνατότητες των Παλαιστινίων, της Παλαιστίνης. Και η ουσία είναι ότι εάν οι Παλαιστίνοι αποδεικνύουν, όπω κατά την άποψή μου συμβαίνει, ότι μπορούν να οικοδομήσουν αυτέ τι δυνατότητε και να λάβουν τη διακυβέρνησή του με πιθανό τρόπο, αυτό δεν είναι μια απάντηση προ το Ισραήλ, δεν αφοπλίζει το Ισραήλ. Σε αυτό θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε έμφαση, ότι υπάρχουν περιοχέ όπου μπορούμε να επιφέρουμε αλλαγέ. Που μπορούν μάλιστα να αποκριθούν σε μέτρα που λαμβάνουν οι Ισραηλινοί. Στην περιοχή Α, όπου οι Ισραηλινοί έχουν τον έλεγχο των μέτρων ασφαλεία και υπήρχαν ακραίε συνθήκε προηγουμένω, δεν θα έπρεπε πλέον να υπάρχουν ανάγκε εφόδων των Ισραηλινών εκεί. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει τρόπο να βοηθήσουμε του Παλαιστινίου ιδιαιτέρως με το δικό μας το έργο, με την αστυνόμευση από πολίτες. Να ολοκληρώσουμε την οικοδόμηση των δυνατοτήτων, ώστε από κάθε μεριά της Παλαιστινιακής Αρχής ο καθένας να μπορεί να κάνει το έργο ασφάλειας και τάξης που απαιτείται. Υπάρχουν και άλλες περιοχές, μεταξύ των οποίων η περιοχή Γάμαση. Ε, και εκεί δίνουμε έμφαση και επικεντρώνουμε την προσοχή μας. Το λέμε στους ανθρώπους ότι η δυτική όχθη ε, είναι χωρισμένη σε τρεις περιοχές, A, B και C. Η Τρίτη περιοχή είναι κατά 60% τα εδάφη της Δυτικής Όχθης και είναι υπό τον έλεγχο του Ισραήλ κατά κύριο λόγο. Οι Παλαιστίνοι κατάφεραν να αναπτύξουν ε, δραστηριότητα στην περιοχή αυτή αλλά χωρί άδεια και την άδεια αυτή, την νόμιμη άδεια πρέπει να την λάβουν ώστε να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε δρόμους οι Παλαιστίνοι για κάποιε πόλει του. Όπω το στεγαστικό πρόγραμμα Wabi που θα είναι η πρώτη πόλη που έχει οικοδομηθεί στην Παλαιστίνη εδώ και πολλά χρόνια, δεκαετίε μπορώ να σα πω. Το πρόγραμμα αυτό, το πρόγραμμα Wahhabi στα βόρεια της Ράμαλα, είναι ένα πρόγραμμα που προβλέπει πολύ καλές οικοδομές, αλλά ήδη υπάρχει διαφιλονικία για έναν δρόμο πρόσβασης οδό πρόσβαση. Είναι πολύ δύσκολο να επιληθεί το σημείο αυτό. Ελπίζουμε ότι θα το πετύχουμε. Αλλά επιμένω, χρειάζεται χρόνο για αυτέ τι λύσει και εμεί τι χρειαζόμαστε τώρα. Τώρα, εάν με αν με ρωτάτε ποιο είναι το αποτέλεσμα του απολογισμού, πρέπει να σα πω για τη Γάζα, για του λόγου που γνωρίζουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και το έχετε ακούσει ξανά και ξανά στο παρελθόν. Τώρα στη Δυτική Όχθη υπάρχει μια ελπίδα ε, οικοδόμησης κρατικών δυνατοτήτων, αλλά πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, πρέπει να επικεντρώσουμε τι προσπάθειε μα σε συγκεκριμένε ενέργειε για να μπορέσουν και οι Παλαιστίνοι να φέρουν ει πέρα στα δικά του έργα και οι Ισραηλινοί να λάβουν αυτά που ελπίζουν και πιστεύουν ότι αξίζουν να λάβουν. Πρόεδρο ευχαριστώ. Εάν συμφωνείτε να ακούσουμε ένα γύρο τριών ερωτημάτων, να έχουμε τρία ερωτήματα κάθε φορά για να μπορέσουν όσο περισσότεροι συνάδελφοι να θέσουν τα ερωτήματά τους. Παρακαλώ, περιοριστείτε σε ένα-ενάμιση λεπτό. Κύριε Ντέβα. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θυμάμαι ότι περάσαμε κάποιο καιρό στο Κοινοβούλιο της Αγγλίας, στο House of Commons και είχατε υποστηρίξει τον John Major στην διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία. Υπάρχει μια χημεία η οποία έχει αναπτυχθεί, η οποία τελικά οδήγησε στον τροματισμό μιας διαμάχης που κράτησε 500 χρόνια. Ακούω λοιπόν τι λέτε, μιλάτε για την οικοδόμηση θεσμών και την ανάπτυξη δυναμικού. Αν δεν υπάρχει όμως η πολιτική εμπιστοσύνη, αν δεν υπάρχει χημεία αν θέλετε, θα κάνετε ό,τι έκανε John Major στην Ιρλανδία. Αν δεν το έχετε λοιπόν εσείς αυτό το κύρος, ποιος θα το κάνει, ποιος θα κάνει τη δουλειά αυτή. Μπορούμε να χορηγούμε τα κονδύλια της Ένωσης στην Παλαιστίνη, αλλά ποιος είναι αυτός ο υπεύθυνος για να δημιουργηθεί αυτή η χημεία, αυτή η εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτικών ηγετών. Ο κύριος Αρσένης. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπλερ έχετε μακρά εμπειρία στην ευρωπαϊκή πολιτική. Και φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλος εμπορικός εταίρος του Ισραήλ. Ωστόσο, οι πολιτικές μας δεν ε, έχουν καταφέρει να επιλύσουν τις διαφορές στην περιοχή. Ποια συγκεκριμένα σφάλματα θεωρείτε ότι κάνουμε εμείς ως Ένωση τα τελευταία χρόνια αν θέλετε μην αποφύγετε την απάντηση στην ερώτηση αυτή και τι αλλαγές θα προτείνατε στις πολιτικές μας αυτές. Και ο κύριος Κάσμαν λέει πρόεδρος. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, καλώς ορίσατε κύριε Μπλερ, καλώς όρισες Τόνι. Μία ερώτηση η οποία είναι παρόμοια αυτή του κυρίου Στέιβενς. Όπως και, είπα, όπως και εσείς είμαι αισιόδοξο από τη φύση μου και θεωρώ ότι θα πρέπει να δώσουμε στον κόσμο την, το δικαίωμα σε υγιεινή άδρευση, πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες και το καθεξής. Αλλά τα πιο πολλά από αυτά δεν τα έχει ο κόσμος εκεί και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει δέσμευση από πλευρά της Παλαιστίνης για την ανάπτυξη της λύσης των δύο κρατών. Δεν είμαστε βέβαιοι όμως ότι αυτό το αποτυπώνει και η δέσμευση του Ισραήλ. Τι μπορείτε να κάνετε λοιπόν από πολιτική άποψη για να αλλάξει η αντίληψη, γιατί όπω ξέρετε οι αντιλήψει και οι νοοτροπίε ε, στην πολιτική είναι πιο σημαντικέ καμιά φορά από τα γεγονότα. Τι μπορείτε να κάνετε λοιπόν προ την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Δύο Βρετανοί συνάδελφοι ανέφεραν τι εμπειρίες μα από τη Βόρεια Ιρλανδία. Με αυτή τη διαδικασία τη βόρεια Ιρλανδία έμαθα κι εγώ ένα-δυο πραγματάκια. Το ένα ήταν ότι τα πράγματα ποτέ δεν είναι τόσο άσχημα ή τόσο όμορφα όσο μοιάζουν να είναι. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν φαίνονται να είναι πολύ αισιόδοξα. Όμως, αν ξεκινήσουν οι, συνομιλίες και οι πρώτες διαπραγματεύσεις, ίσως να βελτιωθεί η κατάσταση. Άσχετα λοιπόν με το τι κάνει κανείς, καθημερινά, η καθημερινή προσπάθεια και η γενικότερη αντίληψή μα είναι ότι κανεί δεν πρέπει να, τα, να το βάζει κάτω σε αυτέ τι περιπτώσει. Δεν πρέπει να τα παρατάει. Ποτέ. Και κάτι ακόμη. Πάντοτε υπάρχει επιλογή. Διότι αν υπήρχε μια συγκέντρωση, λαϊκή συγκέντρωση λόγου χάρη, όλοι όσοι ασχολούνται με το ζήτημα αυτή του στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη έχουν και τι προσωπικέ του ελπίδε, τι προσωπικέ του σκέψει και ιδέε. Τι θα έπρεπε να κάνει κανεί, πώ να προχωρήσει καλύτερα. Η δική μου εμπειρία από τη διαδικασία τη Βόρεια Ιλανδία είναι ότι το να μπορέσει κανεί να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του είναι σημαντικό αλλά πρέπει να είναι και προσεκτικό. γιατί την επόμενη μέρα πρέπει να έχει υπόψη ότι θα ξαναέρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θα ξανασυνεργαστεί με τι δύο πλευρέ. Το δικό μου λοιπόν έργο είναι πρακτικό, καθημερινό. Μιλάμε για καθημερινή άμεση διάδραση με του Παλαιστινίου και του Ισραηλινού, με τι δύο πλευρέ. Η πραγματική μου λοιπόν αντίληψη για το πώ οικοδομείται η εμπιστοσύνη είναι ότι φτιάχνεται μέσω των ενεργειών, τη δράση. Αυτό σα λέω στην ουσία. Μέχρι το 2000 μπορούσε κανείς με τα λόγια να χτίσει την εμπιστοσύνη. Η διαφορά πλέον σήμερα είναι ότι δεν γίνεται αυτό πλέον. Δεν το πιστεύω. Πρέπει να υπάρξουν ενέργειες, δράσεις. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Και ίσω κάποιοι δεν θέλουν να το βλέπουν το θέμα από την προοπτική του Ισραήλ, αλλά να σα το πω. Ε, και εγώ γιατί είναι σημαντικό από την προοπτική του Ισραήλ. Γιατί δεν μπορεί κανεί να το αντιληφθεί αν δεν το δει και από τι δύο πλευρέ το ζήτημα. Λένε ότι πήγαμε στην Γάζα, είχαμε μαζί μα του επίκου μα και τώρα έχουμε την επίθεση τη Χαμά. Ξέρω ότι υπάρχουν επιχειρήματα. Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε εδώ. Αλλά εάν δει κανεί τι συμβαίνει στη Δυτική Όχθη, ε, είναι σαφές ότι παρακολουθούν προσεκτικά τι συμβαίνει σε μια πολύ μικρή έκταση με ανθρώπους που ζουν ο ένας ε, σχεδόν πάνω στον άλλο. Οι Παλαιστίνοι λένε ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ξέρετε ότι θέλουμε τη λύση των δύο κρατών. Τι άλλο θέλετε για να μα δώσετε να βιώσουμε Παλαιστινιακό κράτο. Όμω, ε, μετά όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, η προσπάθεια χτισήματο εμπιστοσύνη έχει διαλυθεί. Μόνο με δράσεις και όχι με λόγια πιστεύω ότι μπορεί αυτό να το ανακτήσουμε. Τι, τι λάθη έχει κάνει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω και δεν ξέρω αν μπορεί να το χαρακτηρίσει κανεί αυτό σφάλμα ή όχι, αλλά αυτή τη συμβουλή την έχω δώσει και στο γεύμα που είχαμε του υπουργού ε, σήμερα. Η Ευρώπη πρέπει να έχει μάλλον την διάθεση να αναλάβει πολιτικό ρόλο εδώ. Είναι σαν να κοιτάζει Ηνωμένε ΗΠΑ και να λέει «Ε, εσείς μπορεί να παίζετε, να παίζετε πολιτικό ρόλο, αλλά επειδή τα χρήματα έρχονται και από εμά, θέλουμε και εμεί μερίδιο σε αυτόν τον πολιτικό ρόλο. Αυτό που έχω να πω λοιπόν εγώ για την πολιτική διάσταση του θέματο είναι ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στο τι κάνουμε πραγματικά και τι μπορούμε να κάνουμε που κανεί άλλο δεν μπορεί να το προσφέρει. Αυτό είναι η πρώτη μα προτεραιότητα. Αυτό θα πρέπει να είναι. Να ενισχύσουμε τους Παλαιστινίου στην οικοδόμηση του κράτους, των θεσμικών οργάνων, των υποδομών τους. Εάν αυτό συμβεί, θα μπορέσουμε να κάνουμε και πολύ περισσότερα. Και θα βρούμε και το άνοιγμα να αναλάβουμε μια πολιτική δράση και ένα πολιτικό ρόλο. Αλλά αν δεν είμαστε καθοριστικοί παράγοντες στην δράση, στις ενέργειες που χτίζουν την εμπιστοσύνη, δεν θα αναλάβουμε τον πολιτικό ρόλο. Και η αντίληψη που υπάρχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται πάρα πολύ από τι δράσει που γίνονται εκεί καθημερινά, λόγω χάρη μέσω τη αστυνόμευση. Η εικόνα αυτή είναι αρκετά καλή ω προ αυτό το θέμα. Και έχει αλλάξει ω προ το παρελθόν. Και μια τελευταία παρατήρηση. Ναι, η αλήθεια είναι ότι παρά τις σημερινές δυσκολίες μπορεί να ξαναξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Αλλά αυτό θα γίνει μόνον εφόσον υπάρξει εμπιστοσύνη. Οι διαπραγματεύσεις τις οποίες θα περάσουν, να είναι αληθινές και όχι απατηλές. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε σημαντικός παράγοντας, αλλά όχι πάντοτε ο πλέον σημαντικός. Κυρία Ντεκάιζερ. Merci. Κύριε Μπλερ, είναι αλήθεια ότι τρέφαν πολλές ελπίδες για την δράση, την πορεία θα μπορούσατε να αναλάβετε εσείς για την Γάζα. Υπήρχαν πάρα πολλά σχέδια για έργα υποδομή, τα οποία δεν μπόρεσαν ίσω να ευοδοθούν. Δεν σα κάνω όμω ερωτήσει για αυτό το θέμα, δεδομένου ότι δεν ήταν και ευνοϊκό το διεθνές κλίμα. Και σήμερα με τον κύριο Ομπάμα και την κυρία Άστον ίσω πάμε πιο μακριά. Υπάρχει όμω ένα σημείο με το οποίο διαφωνώ μαζί σα. Μιλήσατε για την ασφάλεια και αναφέρατε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη το θέμα της ασφάλειας του Ισραήλ και αν ε, κατορθώσουμε να θεσπίσουμε το κράτο δικαίου στην Παλαιστίνη, τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Συμφωνώ μαζί σα ότι όντω είμαστε αλληλέγγυοι στο θέμα τη ασφάλεια του Ισραήλ. Ε, θελήσαμε να είναι και το Ισραήλ και είμαστε υπεύθυνοι για την ασφάλειά του. Αλλά είμαστε ακόμη πιο υπεύθυνοι για την ασφάλεια των Παλαιστινίων. Και αυτό αυτή η διπλή έννοια της ασφάλειας είναι κάτι που θέλω να μας πείτε. Βλέποντας τους αριθμούς, τα τελευταία χρόνια Βλέπουμε δυστυχώς για κάθε θάνατο Ισραηλινού 10 ή 100 θανάτους Παλαιστινίων μηνιαίως. Εγώ τα έλεγξα όλα αυτά τα στοιχεία που σας αναφέρω πάντα καταδικάζαμε αυτά τα οποία γίνονται στο Κοινοβούλιο και τις ρουκέτες και τις τρομοκρατικές πράξεις αλλά και τις εξοδικαστικές δολοφονίες και όλο το θέμα της ασφάλειας των Παλαιστινίων. Όταν θέλουμε λοιπόν να κατανοήσουμε τι ακριβώς γίνεται ένθεν και ένθεν, ποτέ δεν θα πρέπει να μιλούμε για την ασφάλεια του Ισραήλ αν δεν μιλούμε συγχρόνως και για την ασφάλεια των ε, Παλαιστινίων και για την προοδευτική απώλεια των εδαφών τους. Με όλα τα άλλα συμφωνώ. Η κυρία Θεοχάρους. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω ελληνικά, κύριε Μπλερ. Βάλτε ακουστικά εκτός αν καταλαβαίνετε και τα ελληνικά. Παρακολούθησα με πόσο ζήλο υπερασπιστήκατε την απόφαση σας να παρέμβει η Βρετανία στρατιωτικά στο Ιράκ και αναρωτιέμαι αν υπάρχει πολιτικός τρόπος πολιτικά μέσα να ανακοπεί το έγκλημα του επικισμού το οποίο επιτελεί αυτή τη στιγμή το Ισραήλ καθώς επίσης και αν υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί η καταστροφή της οποιασδήποτε βασικής υποδομής. Είπατε ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εκ των κάτω προς τα πάνω ένα Παλαιστινιακό κράτος. Αλλά όταν βλέπουμε ότι μόλις δημιουργηθεί μια βασική υποδομή είτε στη Γάζα είτε σε πόλεις της Δυτικής Όχθης αμέσως η πολεμική μηχανή του Ισραήλ βρίσκει μια αφορμή και τα καταστρέφει όλα και τα ισοπεδώνει. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάποιος τρόπος για να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Όσον αφορά τον επικισμό, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι ο επικισμός είναι ένα έγκλημα πολέμου το οποίο πάντοτε υπονομεύει και ναρκοθετεί οποιαδήποτε προσπάθεια λύσης και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι με απόφαση του Βρετανικού εφετείου ένα άλλο έγκλημα επικισμού που έγινε σε μια γειτονική προς την Παλαιστίνη χώρα έχει, έχουν καταδικαστεί όλες οι συνέπειες αυτού του εγκλήματος και εκεί δεν έκανε τίποτα η Βρετανία για να ανακόψει αυτό το έγκλημα. Μήπως θα πρέπει να κάνουμε κάτι προς την κατεύθυνση της Μέσης Ανατολής αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ. Καλώ Welcome from Καλώς όρισες, Τόνι, και εγώ δεν θα ρωτήσω τίποτα για την Γάζα. Βεβαίως καταδικάζουμε την απώλεια ζωών του αμάχου πληθυσμού και από τις δύο πλευράς. Αλλά Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για, την, ε, για το πρόβλημα της λειψιδρίας. Από ό,τι ξέρουμε, μόνο 5% των υδάτων είναι πόσιμα. Μπορείς να μας πεις πώς βλέπεις το θέμα αυτό. Είπε στην προηγούμενη Παρασκευή ότι είσαι υπέρ της ε, δημιουργίας της Παλαιστίνης και πώς πιστεύει εσύ ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Λωρίδα τη Γάζα είναι κάτι το οποίο υπομονεύει τι προσπάθειε. έχοντας εσύ την εμπειρία της Ιρλανδίας βλέποντας πώς η Χαμάς συνεργάζεται με τους τρομοκράτες πιστεύεις ότι η Χαμάς μπορεί να ακολουθήσει έναν δρόμο που θα τη φέρει στη δημοκρατία και στην ειρήνη uh, First of all, uh, in recent... Ε, ευρύτατα ερωτήματα. Για το θέμα της ασφάλειας και κατά πόσο είναι ζήτημα και των Παλαιστινίων όσο και των Ισραηλινών. Βεβαίως και είναι. Όμως τελικά η ασφάλεια και το πώς θα την ανισχύσουμε κατευθείαν διοχετεύεται και στην προσπάθεια την ειρηνευτική. Ένας από τους λόγους λοιπόν που είναι τόσο σοβαρό να ενισχύσουμε τις δυνατότητες των Παλαιστινίων για, την, για το κράτος δικαίου και για να επικρατήσει ασφάλεια είναι ότι όπως είπε και ο πρόεδρος των Παλαιστινίων και λέει θέλουμε με ένα νόμο, ένα όπλο, μία αρχή. Δηλαδή να υπάρχει μία Παλαιστινιακή αρχή που να διαθέτει τα μέσα να επιβάλλει το κράτος δικαίου. Την τάξη. Και εάν θέλουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα πρέπει να δούμε τις διαφορετικές του πτυχές από τη σωστή προοπτική. Πολλοί Παλαιστίνοι από την ε, Λωρίδα της Γάζας βλέπουν τι έχει γίνει λόγω χάρη στη Δυτική Όχθη, στην Ιερουσαλήμ. Βεβαίω βλέπουν ότι έχουν γίνει παράνομε ενέργειε κατά τη Παλαιστινική Αρχή. Ο καθένα θα έχει επιχειρήματα υπέρ και κατά. Όμω η ασφάλεια, η κατάσταση ασφάλεια είναι μια δυνατότητα λύση. Και η οικοδόμηση δυνατοτήτων είναι τόσο σημαντική για του Παλαιστινίου, διότι λόγω χάρη, όπω συνέβη πριν από λίγου μήνε, Εάν υπάρξει κάποιο ξέσπασμα βίαιων γεγονότων μεταξύ δύο συμμοριών ας πούμε, που έγινε στην Παλαιστινιακή περιοχή, θα πρέπει να μπορεί η Παλαιστινική Αρχή να καταστήλει τέτοιου είδου δράσει. Αυτό λοιπόν είναι τεράστια σημασία. Μέρο τη σοβαρότητα του ζητήματο είναι ότι κάποιοι δεν θέλουν να τα σκέφτονται αυτά. Βλέπουν μόνο τι συνόδου κορυφή, τι διαπραγματεύσει και ούτω καθεξή. Όχι αυτά τα ζητήματα είναι στην καρδιά του προβλήματος, τα θέματα της ασφάλειας. Διότι διαφορετικά και αν συνεχιστεί η σύγκρουση, η έλλειψη ισορροπίας στην, στην εξουσία θα συνεχιστεί και ανησυχητικοί αριθμοί θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Άρα η λύση και η ειρήνη είναι να έρθουμε σε ειρηνευτικές διαδικασίες με του προσώπους τη Παλαιστινική Αρχή που να διασφαλίζουν την τάξη εκεί τώρα για την κατοχή. Η κατοχή Βεβαίω, δημιουργεί το εξή πρόβλημα. Δεν είναι μόνο οι περιορισμοί για την ζωή των Παλαιστινίων το πρόβλημα. Είναι ότι είναι δύσκολο και η οικονομία των Παλαιστινίων να αναπτυχθεί με τόσους περιορισμούς να λειτουργούν. Όμως η πραγματικότητα είναι η εξή, ότι θα έρθουν οι περιορισμοί μόνο να έχουν επαρκεί δυνατότητε μόνο του να εξασφαλίσουν την ασφάλεια και την τάξη. Αυτό το συζητήσαμε και το συζητάμε εντόνω τις τελευταίες ημέρες και έχουμε πολλά επιχειρήματα υπέρ του δικού μας, ε, της δικής μας θεώρησης. Πρέπει να έρθει κανείς και να επισκεφτεί την περιοχή για να δει τι γίνεται στην Ιεριχώ, στη Ράμαλα, στη Βιθλεέμ, στην Άμπλους και αλλού. Εκεί υπάρχουν κάποιες ε, δυνατότητες να βρεθεί απάντηση. Δεν είναι η καλύτερη η ιδανική λύση, αλλά είναι ο μόνος τρόπος να προχωρήσουμε. Και Ήδη έχουμε κάποια προγράμματα οικοδόμηση, ε, κάποια υλικά. Έχουμε λάβει τι άδειε για να τα φέρουμε ε, στην ε, περιοχή των κατεχομένων. Θα γίνουν και οι διαγωνισμοί, θα οικοδομηθούν τα προγράμματα, αλλά χρειάζεται ο απαραίτητο εξοπλισμό. Εδώ έχουμε αγώνα με το χρόνο και θα πρέπει οι Ισραηλινοί να χαλαρώσουν την πολιορκία του για να μπορέσουν να δίνουν τα απαραίτητα έργα. Και σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό, την υδροδότηση θα συνεχίσουμε να κάνουμε τις ίδιες προσπάθειες όπου κάναμε και στο παρελθόν και όσο αφορά τη Χαμάς. Κοιτάξτε, δεν αφιβάλλω σε καμία περίπτωση ότι εάν υπάρξει ένας ε, σοβαρός ρυθμός, σταθερός ρυθμός με ρεαλιστικές προοπτικές ειρήνευσης, τότε η Χαμάς θα έχει και μια επιπλέον επιλογή που θα είναι και η σωστή επιλογή που θα μπορέσει να κάνει. Δηλαδή, ή θα συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία ή θα βγει εκτό παιχνιδιού. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων στη Γάζα, εάν δουν να υπάρξουν ρεαλιστικέ προοπτικέ βιώσιμου Παλαιστινικού κράτου, θα ε, δεχτούν τη λύση των δύο κρατών. Αυτό είναι η ελπίδα όλων. Ότι ο λαό, οι άνθρωποι με του οποίου μιλώ στη Γάζα συνεχώ, είναι πεπισμένοι για αυτό το ενδεχόμενο. Τώρα, κάποια στοιχεία της Χαμάς η αρχή του κουαρτέτου δεν είναι να έχουμε συνομιλίε με την ε, Χαμά, αλλά συναντούμε ανθρώπου. Δεν υπάρχει λοιπόν εδώ κενό στην επικοινωνία μα. Μεν. Αλλά εάν υπάρχει δυνατότητα να λάβει κανεί απόφαση, θα είναι πιο εύκολο να λάβει τη σωστή απόφαση αν υπάρχουν επιλογέ στην ερευνητική διαδικασία. Κύριε Μπλερ, είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ ιδιωτικά το Ισραήλ και την Δυτική Όχθη πριν από τρει εβδομάδε περίπου και πρέπει να πω ότι δεν ε, συμμετέχω. Δεν, είμαι, δεν συμφωνώ με την αισιοδοξία σας με την επίσκεψη αυτό, αυτή, γιατί βλέπουμε ότι η Βυτική Όχθη έχει καταντήσει ελβετικό τυρί από τις τρύπε. Και επιπλέον βλέπω, βλέπουμε ότι πρόσφατα όταν ο Τζο Μπάιντεν επισκέφθηκε την Ιερουσαλήμ βλέπουμε πως οι Ισραηλινοί ανακοίνωσαν τις ε, δραστηριότητες ε, επικισμών στη Βετική Όχθη. Αυτό φυσικά δεν βοηθάει στην δικοδόμηση εμπιστοσύνης και φυσικά ξέρουμε τις τηλεφωνιακές επικοινωνίες μεταξύ Νιτανιάου και, και Μέρκελ. Όλα αυτά με οδηγούν να πιστέψω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να είμαστε αισιόδοξοι. Είχα έναν πολύ νέον Ισραηλινό οδηγό και τον ρώτησα γιατί δεν έχει υποδεχτεί η Παλαιστίνη τη λύση των δύο κρατών ήδη. Δεν έχει τελειώσει ο χρόνος. Και ο Ισραηλινός μου απάντησε ότι τελειώνει ο χρόνος όχι για τους Παλαιστινίους αλλά για μας. Τι εννοείς τον ρώτησα. Ότι οι Παλαιστινοί κάποια μέρα δεν θα ζητήσουν λύση δύο κρατών αλλά ενός κράτους με ίσα δικαιώματα για τους Παλαιστινίους και αυτό θα το τέλος για το κράτος του Ισραήλ. Και το Ισραήλ φυσικά δεν τους δίνει τα δικαιώματα αυτά για να μην δημιουργηθεί μια κατάσταση apartheid. Πώς ε, τοποθετήσετε εσείς έναντι της τοποθέτησης αυτής και κατά δεύτερον, γιατί να μην ακολουθήσουμε τη διαδικασία Dayton, να καλέσουμε τις δύο πλευρές και να πούμε ότι δεν θα φύγετε από εδώ μέχρι να βρεθεί μια λύση. Ο Μιλόσεβιτς δεν, θέλησε να υπογράψει, δεν ήθελε να υπογράψει την λύση αυτή, αλλά τελικά την υπέγραψε. Γιατί να μην ακολουθήσουμε λοιπόν την ίδια, την ίδια προσέγγιση. Κύριε Χατζηγεωργίου. Κύριε Μπλερ, να σας καλωσορίσω και εγώ στη συνεδρία μας Είμαι της άποψης ότι μετά από τόσα πολλά χρόνια πολύ απίστευτης τραγωδίας του Παλαιστινιακού λαού πρέπει κανείς να πει το σαφές ότι η διπλωματία πρέπει να, πρέπει να έχει τελειώσει. Πρέπει να περάσει κανείς σε πράξεις. Θα είμαι έτσι λίγο εχμηρός μαζί σας, λέγοντας σας ότι είστε ένας κατεξοχήν διπλωμάτης αλλά έχοντας κατά νου ότι η δουλειά της διπλωματίας θα πρέπει να έχει τερματίσει τη δραστηριότητά της, νομίζω ότι πρέπει να σας στείλει το μήνυμα ότι πρέπει να εργαστούμε προς την κατεύθυνση των πράξεων. Εσείς είστε ο άνθρωπος ο οποίος έστειλε βρετανικά στρατεύματα στο Ιράκ για να βρουν μία μπουκάλα με χημικά. Και δείχνετε τώρα μια εικόνα, επιτρέψτε μου να πω, απλώς επικοινωνιακή και διπλωματική, απέναντι σε ένα πρόβλημα που δεν αντέχει πια στο χρόνο. Θα σας στεναχωρήσω αν σας πω ότι πιστεύω ότι δεν θα πετύχετε. Και βάλτε αν θέλετε εσείς μόνο σας ένα ορόσημο χρονικό. Πότε θα πείτε ότι κλείνει αυτή η προσπάθεια και δεν έχει καταλήξει παρά μόνο αρνητικά. Δίνετε στον εαυτό σας ακόμα ένα χρόνο, δυο, πέντε, πρέπει επιτέλους να αποφασίσει η διεθνής κοινότητα και εμείς εδώ είμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι χωρίς κυρώσεις προς το Ισραήλ δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Κύριε Στάνοκ, ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Μπλερ, είστε ειδικό απεσταλμένο Η Ρωσία είναι ένα από τα αφεντικά σα στο κουαρτέτο, αλλά πρόσφατα είπε ότι ο αγωγός που έτσι θα μπορούσε να χρησιμεύσει και θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για το Ισραήλ και απειλή μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας για κυρώσεις και κατά τον πόλεμο στο Λίβανο ανακαλύφθηκαν ρωσικά πυρομαχικά στη Χεσμπολά. Θεωρείται ότι κάνει αρκετά η Ρωσία για να μας πείσει, να πείσει το Ισραήλ για τις ειρηνικές της προθέσεις και κατά δεύτερον Υπάρχουν ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις στην Παλαιστίνη και ξέρουμε ότι πολλές από αυτές έχουν συμπεριληφθεί σε κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων, όπως η πολλά, ο Πιλ Νιούτον εδώ είμαι. Η Βόρεια Ιρλανδία αναφέρεται ως παράδειγμα και ο Τζον Χιούμ, ο οποίος είχε κερδίσει το βραβείο Ειρήνης ε, για τη διαδικασία αυτή, μου είχε εξηγήσει ότι είχε εξηγήσει στον Τζέρι Άντεμ στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα περί ίσων δικαιωμάτων, το όφελος και φυσικά το θετικό ήταν ότι και η Βόρεια Ιρλανδία και η Ευρωπαϊκή και το Βασίλειο ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν ισχύει όμως ε, για τη Μέση Ανατολή. Μπορούμε να πούμε όμως στην Ισραήλ και στην Παλαιστίνη να ξεχάσουν τη θρησκεία, να ξεχάσουν τη θρησκεία και να μιλήσουν μόνο για τα ίσα δικαιώματα. Αυτό πιστεύετε ότι ενδεχομένως θα βοηθούσε? Yeah, well, the Πολλές ερωτήσεις ενδιαφέρουσες. Χαίρομαι που άκουσα ότι εξήγησε ο Τζον Χιούμ στον Τζέρι Άνταμς τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν είχα και ένα αντίγραφο να το δω κι εγώ, θα μπορούσα να το πάρω μαζί μου να τον κόσμο και να εξυπηρετήσει κι άλλους. Τέλος πάντων. Σε σχέση με την Δυτική Όχθη, εάν πείτε σε κάποιον ότι δεν συμβαίνει τίποτε καλό στη δικαιοχθάντη, θα σας πούνε ότι είστε απεσιόδοξο. Αν σα πούνε ότι κάτι καλό συμβαίνει, θα σας πούνε είστε υπεραισιόδοξο. Τι έχω να πω εγώ για την προσέγγιση με τη Δυτική Όχθη. Εάν δείτε τη ζωή στι μεγαλύτερε Παλαιστινιακέ πόλει σε σχέση με το τι συνέβαινε πριν από δύο χρόνια, τα πράγματα βελτιώθηκαν. Και βεβαίω αυτό δεν σημαίνει ότι ακόμη πρέπει να διανυθεί πάρα πολύ μεγάλο δρόμο. Τώρα, σε σχέση με το ένα κράτος, τη λύση ενός κράτους. Ακούω και τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους να μιλούν για αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα. Δεν μπορώ να δω πώς μπορεί να διευθυνθεί μια τέτοια κατάσταση, να κυβερνηθεί ένα τέτοιο ένα κράτος. Ο τρόπος για τον οποίο έφτασε ο κόσμος σε αυτή τη λύση των δύο κρατών δεν είναι διότι όπως συνήθως συμβαίνει υπάρχει πίεση, αλλά διότι με όλη τη λογική που χρησιμοποίησαν είδε ότι δεν υπήρχε άλλη λύση. Δεδομένου ότι υπάρχει ε, η, λαός Ισραηλινός και λαός Παλαιστινίων. Θέλουν λοιπόν οι Παλαιστίνοι να έχουν ε, για λόγους αξιοπρέπειας ένα κράτος και οι Ισραηλινοί κατέχουν ένα μέρος των εδαφών των Παλαιστινίων. Εάν κάποιος εκφράζεται υπέρ αυτής της λύσης, σημαίνει ότι είναι πολύ αποκεντρωμένος από την κατάσταση υποκριτία. Δεν είναι λύση. Τώρα, κάποιο άλλο συνάδελφο είπε η διπλωματία να αντικατασταθεί με ενέργειες, με δράσεις. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι, αυτός είναι ο κατάλληλος δρόμος. Καλύτερα μέτρια διπλωματία παρά ε, μη διπλωματία καθόλου. Τώρα, σε σχέση με το Ιράν και τη Ρωσία. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες της μη κυβερνητική οργάνωσης στην οποία αναφέρεστε. Το θέμα της Ρωσίας και του Ιράν είναι θέμα διαπραγμάτευσης μεταξύ των Ιρανών, των Αμερικανών και πρέπει να πω σε σχέση με τη δουλειά τη δική μου και όταν ανέλαβα εγώ εκ μέρους του κουαρτέτου ότι αυτή η οικογένεια δεν είναι και ότι πιο αρμονικό υπάρχει ως αρχηγός αλλά εγώ κάνω τη δουλειά με σοβαρότητα. Τώρα, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η... Ένα μέρος της λύσης είναι στην περιφερειακή προσέγγιση. Αλλά αυτό σημαίνει ότι συγχρόνως θα προχωρήσει και η ε, ειρηνευτική διαδικασία. Το ένα δεν μπορεί να γίνει χωρίς τον άλλο. Όταν ε, τέθηκε σε κίνηση η όλη διαδικασία το 2002 ήταν η κατάλληλη στιγμή. Και αυτό το λέω στους Ισραηλινούς, ότι υπήρχε, αυτό ήταν ένα σημαντικό άλμα προς τον πώς για τον αραβικό κόσμο. Μην παραγνωρίσετε λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία για την ειρήνη πρόκειται για κάτι το νόμιμο. Είναι ένα επιχείρημα το οποίο πρέπει να χρησιμοποιεί στι ε, διαπραγματεύσει. Αλλά έχω την εντύπωση ότι οι πραγματικές διαπραγματεύσεις με πολιτικό περιεχόμενο θα είναι πολύ δύσκολο να προβάλλουν πρώτα την περιφερειακή ε, διάσταση. Και αλλά αν μπορέσουμε να το καταθέσουμε, όντως για μένα πρόκειται για μια διάσταση πάρα πολύ σημαντική. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος της συνεδρίασής μας. Πιστεύω ότι ήταν εξαιρετικά χρήσιμη και ενδιαφέρουσα η συνάντηση του σημερινού απογεύματος. Θα ήθελα να πω σε όλα τα μέλη των κοινοβουλευτικών επιτροπών που συμμετείχαν και στους διερμηνείς καθώς και στον ειδικό μας προσκεκλημένο τον κύριο Μπλερ ότι τον ευχαριστούμε διότι μοιράστηκε την εμπειρία του και την απόψη, του με εμάς.